Okay, good morning. I think we can start uh, the meeting of the subcommittee on human rights. Καλημέρα, ας ξεκινήσει η συνεδρίασή μας. Σας εγκρίνουμε πρώτα απ' όλα την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχει κανεί αντίρρηση, εγκρίνεται. Μετά θα ήθελα να κάνω κάποιε ανακοινώσει τη Προέδρου. Χτες, πολλοί από εμάς, δηλαδή η κυρία Ροχμπίλερ Κούκαν και εγώ, πήγαμε επιτέλους στο Συμβούλιο να μελετήσουμε το έγγραφο το οποίο είναι η αξιολόγηση του διαλόγου με την Κίνα. Θα θυμάστε πως παλέψαμε για να έχουμε περισσότερη πρόσβαση στις πληροφορίες για να μπορούμε να μειχθούμε στα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, και ήταν κάπως ε, διασκεδαστικό να πάμε στο Συμβούλιο για να επιτηρήσουμε για να δούμε ένα έγγραφο με κάποιον πάνω από το κεφάλι μας και δεν μπορούσαμε να το πάρουμε μαζί μας είναι ένα βήμα σε μια διαδικασία στην οποία τελικά θα αποκτήσουμε πρόσβαση και ίσως στο μέλλον να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε σε ένα δωμάτιο στο Συμβούλιο. λοιπόν, άξιζε τον κόπο. Οπότε δεν μου επιτρέπετε να πω και τίποτα για το έγγραφο αλλά κάτι έμαθα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα γιατί ο διάλογος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την Κίνα έγινε πράγματι και θα γίνει μια ενημέρωση στις 15 Ιουλίου τελευταία συνεδρία πριν διακόψουμε. Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά την απόφαση του διευρυμένου Προεδρείου να στείλει μια μικρή αντιπροσωπεία στον Μπεσλάν, στη Ρωσία, για να τιμήσουμε την τραγωδία του Μπεσλάν. Είναι η εκτεπέτειο την 1η Σεπτεμβρίου της ε, τρομοκρατικής επίθεσης που τερμάτισε με δραματικό τρόπο τερματίστηκε με δραματικό τρόπο αυτή η πολιορκία και πάνω από 100 παιδιά έφυσαν τις ζωές τους. Μια εθνική τραγωδία και μαζί με την Αντιπρόεδρο Ανδρικιένη και την συνάδελφο τον κύριο Μπέρμαν θα πάμε. Μας προσκάλεσαν ε, τοπικές υπερφυριακές ΜΚΟ. Η τρίτη μου ανακοίνωση αφορά τα κατεπήγοντα και την διαδικασία. Υπάρχει μια επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών, την οποία έχω υπογράψει εγώ ως πρόεδρος Υποεπιτροπής Δικαιωμάτων και τον πρόεδρο της διάσκεψης των πρόεδρων των Αντιπροσωπείων. και εκεί πέρα προτείνουμε το διευρυμένο Προεδρείο της Επιτροπής Εξωτερικών να συζητήσει διαδικασία του κατεπήγοντος και το πώς θα μπορέσουμε εμείς να αναμειχθούμε πιο πολύ στην επιλογή θεμάτων για την διαδικασία αυτή. Γιατί πολύ συχνά προκύπτουν αυτά τα θέματα από συζητήσεις και ακροάσεις και άλλες εδώ πέρα συνεννοήσεις και φυσιολογικό είναι να έχουμε κάποιο ρόλο στη διαδικασία. Κατόπιν παρόλες τις ε, παρεμβάσεις ε, στην Συρία τι συνέβη ο Αλχασάνη που έχει λάβει το βραβείο Μάρτιν Έναλς για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 2010 καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών και αυτό το αναφέρω γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε θέσει ένα ψήφισμα το Σεπτέμβρη και καλούσε τις ε, Συριακές Αρχές να απελευθερώσουν τον κύριο Αλχασάνη αμέσως. Και είναι πράγματι λυπηρό και ανησυχητικό να διαβάζουμε το πώς ε, καταδικάστηκε. Κατηγορήθηκε γιατί θεωρήθηκε πως υποσκάπτει το ηθικό του έθνους και επίσης για διασπορά ψευδών ειδήσεων και δικάστηκε και κλεισμένο των θυρών χωρίς δικηγόρο. Τέλος, ο Μουχανάνταλ Χασάνη καταδικάστηκε και με βάση κάποια άρθρα του ποινικού κώδικα. Και είναι προφανές τώρα πως η διαδικασία αυτή δεν εκπληρώνει κανέναν όρο της δικαιιστικής. Όπως λένε πολλοί διακεκριμένοι δικηγόροι και το Ευρωμισογειακό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συνεχίζουμε βέβαια να ζητάμε την άμεση απελευθέρωσή του. Κατόπιν, καλωσορίζω την απελευθέρωση του κυρίου Μακπάκη Ιρανού δημοσιογράφου στις 23 Ιουνίου ο οποίος είναι ιδρυτής της ε, εταιρείας για τις υπεράσπισης ε, των ε, δικαιωμάτων των φυλακισμένων και αυτός έλαβε το βραβείο Μάρκ Νένταλ στο 2008. Ο Μαρτ Μπάκη συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2008 σε ένα κύμα συλλήψεων διαδηλωτών και παραμένει Βεβαίω ε, εξακολουθεί να είναι κατηγορούμενος για προπαγάνδα κατά του Ισλαμικού κράτους και εμεί ζητούμε να αποσυρθούν αυτές οι κατηγορίες. Τώρα, συνάδελφοι, θα ήθελα να δούμε το σημείο 3 μερίσια διάταξη που αφορά την επίσκεψή της αντιπροσωπείας μας στην Ουάσιγκτον. μόλις έρχεται και η κυρία Γκάλ βλέπω οπότε τα βασικά εν πάση περιπτώσει αποτελέσματα θα μπορούσα να σα τα παρουσιάσω και εγώ και ελπίζω η κυρία Γκάλ να εξηγήσει τι έμαθε εκεί στην Ουάσιγκτον και ίσως δεν ξέρω θα θέλατε να δείτε και κάποιες φωτογραφίες εκεί από την επίσκεψή μας εδώ είναι η αντιπροσωπεία στο Κογκρέσο uh, uh, μαζί με μέρη εκεί πέρα, μέλη του Κογκρέσου τα δύο τους πρόεδρους της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ Είμαστε σε μια δεξίωση. Σε μια δεξίωση του Freedom House που ήταν πολύ φιλόξενοι και μας μίλησαν και όλα αυτά. Και αισθανθήκαν πως υπάρχει έτσι μια υπερατλαντική σχέση με τις ΜΚΟ. <laughs> Εδώ βλέπετε τον κύριο Χάρις με δύο πολύ όμορφες παρουσίες. Και βλέπετε εκεί πέρα και τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Στην άλλη μεριά πάλι της τράπεζας στο Κογκρέσο. Κάτι λίγο πίσω στην προηγούμενη κονίτσα. Ευχαριστώ. Θα αναφέρω εδώ τους συναδέλφους. Από τα αριστερά βλέπετε την Άννα Γκόμες, μετά τον Λάζλο Τούκες, εμένα, η οποία Μαρίτε δυστυχώς ε, δεν μπορεί να παραστεί, έχει ανηλυμένη υποχρέωση. Και άλλες εικονίτσες λοιπόν. Να σας πω τώρα τα βασικά. Πολλές από τις συζητήσεις μας αφορούσαν ε, το κλείσιμο του Γουαντανάμο και εδώ δυστυχώς από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση Ομπάμα δεν καταφέρνει να προχωρήσει όσο γρήγορα θα ελπίζαμε εμείς ε, στην Ευρώπη. Οπότε η σύσταση είναι να το παρακολουθήσουμε αυτό το ζήτημα και βεβαίως ε, να συζητήσουμε πώς μπορούν να βοηθήσουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με το να υιοθετήσουν κρατούμενους του Γαντανάμου που δεν κατηγορούνται για τίποτα. Και ταυτόχρονα να τονίσουμε στις συζητήσεις την ανάγκη συμμετοχής ε, σε συζητήσεις για την πολιτική κράτηση στον ΗΠΑ, γιατί όπως ξέρουμε ε, δεν ε, εκπληρώνει αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε δικαιώματα των ε, κρατουμένων και κατηγορουμένων και είχαμε πρόσφατα ανησυχητικές περιπτώσεις όπου φαίνεται πως η ΕΠΑ θα συνεχίσει να κρατεί κρατουμένους χωρίς ε, κατηγορία, χωρίς ε, πιθανότητα δίκης. Αυτό το είπαμε σε όλες μας συζητήσεις, πως δεν είναι αποδεκτό από εμάς. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι πως ε, η προώθηση της δημοκρατίας ίσως έχει περάσει σε μια νέα φάση γιατί η κυβέρνηση Ομπάμα δεν έχει το ίδιο βάρος που θα είχε ίσως ε, η κυβέρνηση Μπούς στο να προωθεί τη δημοκρατία σε άλλες χώρες και συμφωνήσαμε πως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε εδώ ε, μια εκδήλωση για την προώθηση της δημοκρατίας με τις οργανώσεις ε, τις αμερικανικές ε, που προωθούν τη δημοκρατία. Οπότε ελπίζω οι Αμερικανοί φίλοι μας ε, από αυτές τις οργανώσεις να έρθουν εδώ. Επίσης, πολλοί θεωρήσαμε πως υπάρχει ανάγκη να συζητήσουμε πώς θα προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα τη δημοκρατία και αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις για νέα μέσα. Έχουμε το γνωστό μέσο βεβαίως που γνωρίζετε όλοι, αλλά κάποιοι θεωρούν πως ε, δεν εκπληρώνει ίσως ε, τις απαιτήσει εκείνες που είναι έτσι άμεσες. Μια, κάτι το οποίο είχαμε σκεφτεί και θα μπορούσατε ίσως να αποφασίσετε είναι σε μία από τις ε, προσεχείς εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας να αφορά την ε, προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μετά είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις για το διάλογο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φαίνεται πως πρέπει να μιλήσουμε με τους Αμερικάνους για το τι είναι επιτυχής τέτοιος διάλογος, πώς πρέπει να γίνεται και ποιες είναι οι εμπειρίες μας από διάφορες χώρες. Οπότε συζητήσαμε αρκετές εμπειρίες στον διάλογο με την Κίνα, τη Ρωσία και με άλλες χώρες. Φαίνεται πως έχουμε παρόμοιους στόχους, οπότε θα πρέπει να συγκρινούμε τις εμπειρίες μας. Και τέλος θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε ως μέλη της Υποεπιτροπής να έρθουμε σε επαφή και να αποκτήσουμε μια σχέση με μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάποιες κοινέ δηλώσεις επιλεκτικά για επίκαιρα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό το οποίο θα ήταν πολύ ενδιαφέρον θα ήταν να γίνει μια συνεδρίαση σχετικά στο πλαίσιο του διατλαντικού διαλόγου βουλευτών και πολλά μέλη της υποεπιτροπής ε, είναι αναμειγμένες σε αυτό το διάλογο. Οπότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μαζί τους για το πώς θα γίνει αυτό. Αλλά οπωσδήποτε υπήρχε ένα ενδιαφέρον μεταξύ των βουλευτών εκείνων που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα για τη συνεργασία. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Κυρία Γκάλ, λοιπόν, ελπίζω να θέλετε να πείτε κάποια πραγματάκια για την Ουάσιγκτον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είπατε τα πάντα. Δεν θα μπω πλέον σε λεπτομέρειες. Η παρουσίαση που έγινε είναι αρκετά πλήρης και το γραπτοκείμενο επίσης. Να υπογραμμίσω όμως τρία θέματα. Καταρχάς κάτι το οποίο αναφέρατε ήδη, αλλά το οποίο είναι ένα από, τα πιο σημαντικ... από τις πιο σημαντικές εντυπώσεις που αποκτήσαμε εκεί. Είναι καλό το να λέει κανείς ότι υπάρχουν κάποια όργανα τα οποία προσπαθούν να προωθήσουν τη δημοκρατία και ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είναι επίσης σημαντικό να έχει κανείς την δυνατότητα να ε, βοηθήσει οικονομικά τις οργανώσεις αυτές με ταχύτητα και σε χρόνο γενικά έφετο έτσι ώστε να μπορούν να αντιδράσουν έγκαιρα. Αυτά τα όργανα με τα οποία συναντηθήκαμε νομίζω κάνουν, κα... κάνουν πολύ καλή δουλειά και θα πρέπει να δούμε ε, πώς εμείς μπορούμε να βελτιώσουμε τις δικές μας διαδικασίες για να τα χρησιμοποιούμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Από την άλλη πράγματι υπάρχει περαιτέρω ανάγκη διαλόγου και θα πρέπει να το υπογραμμίζουμε αυτό όλο περισσότερο. Είναι σαφές ότι και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτόν τον νομοθετικό σε εισαγωγικά διάλογο, σε διάλογο δηλαδή ανάμεσα στα δύο νομοθετικά σώματα. Τώρα, οι εντυπώσεις μου από αυτές τις συναντήσεις νομίζω ότι ήταν χρήσιμες. Έχει ενδιαφέρον να διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο διαιρεί, αν θέλετε, το Κογκρέσο και το State Department και έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε επαφές και δύο και ε, με τις δύο αυτές, ε, με τους δύο αυτούς θεσμούς. Είναι σαφές ότι όπως και ο πρέβης Ντάμφιλ μας είπε χρειάζονται την ανάγκη μας και από ό,τι καταλάβαμε από αυτά τα οποία μας είπε πράγματι η Αμερικανική κυβέρνηση θέλει να κλείσει τον Γκουαντάναμο αλλά χρειάζεται βοήθεια για να το κάνει αυτό. Αυτό είναι σαφές πλέον. και έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς τα θέματα της εμπλοκής, της πολιτικής εμπλοκής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εξελιχθούν στο μέλλον. Σαν υποεπιτροπή, ανεξάρτητα από ε, το σε τι κατάσταση βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι καθήκον μας να προσπαθήσουμε να προκαλούμε αυτήν την πολιτική εμπλοκή όπου αυτό είναι χρήσιμο. Και αυτό θα πρέπει να γίνει αισθητό και στη Washington. Ευχαριστώ Κίνγκα Γκάλ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποια παρατήρηση να κάνετε, δεν νομίζω. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω Είπαμε ότι ίσως θα πρέπει να προωθήσουμε και το Φόρουμ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, να το βοηθήσουμε. Φυσικά αυτό θα πρέπει να το κρίνουν πρώτα οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις αν είναι απαραίτητο. Αλλά υπάρχει ένα τέτοιο φόρουμ ας πούμε με την Κίνα, ένα σεμινάριο πάντως. Ε, νομίζω ότι αντίστοιχες ε, ρυθμίσεις μπορούμε να κάνουμε και με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο διάλογός μας με τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι διαφορετικής φύσεως, αλλά υπάρχει πράγματι μεγάλη σύγκληση και συνδυασμός απόψεων ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ακόμα καλύτερα τις δυνατότητες τις οποίες μας παρέχει η κυβέρνηση Ομπάμα. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και θα ήθελα να περάσω στο σημείο 4 ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μισελ Τίλεμανς, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΚΟΧΟΜ στην υπηρεσία της ΥΠΑ του εκπροσώπου. Είναι μια καινούργια κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί. Εδώ πάντα είχαμε εκπροσώπους των προεδριών. Υπογραμμίστηκε όμως ότι ο κύριος Τίλεμανς δεν είναι εδώ σαν εκπρόσωπος της Βελγικής Προεδρίας. Αλλά πρόεδρος Κόχομ στην υπηρεσία της υπάτης εκπροσώπου. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με μια σημαντική αλλαγή και μένει να δούμε αν α, τελευταίος μισός χρόνος ήταν διαφορετικός από αυτούς που προηγήθηκαν. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Η συμφωνία για το EIS έχει ήδη υπάρξει. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν νέες δομές στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι η συμφωνία στην οποία έχουμε καταλήξει ήταν σημαντική για όλους. Έχει συμφωνηθεί ότι στο κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο στρατηγίου αυτής της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης θα υπάρχει και μια σαφέστατη ισχυρή δομή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Βαρόνια Άστον η ίδια το υπογράμμισε αυτό και είπε ότι ε, θέλει να υπάρχει ένα σύνδεσμος ο οποίος ε, να ενώνει και μέσα από τα ανθρώπινα δικαιώματα όλες τις δομές που ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει υπογραμμίσει επίσης ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσουν να δουλεύουν τα πράγματα και όταν συναντηθήκαμε εδώ και 15 μέρες μας είπε ότι θέλει να συζητήσει μαζί μας πώς θα οργανωθεί το Προεδρείο του Κόχομ. Και γι' αυτό με χαρά βλέπω ότι η Βελγική Προεδρία υποστηρίζει το ότι αυτή η προσπάθεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να βασιστεί στα κεντρικά στις Βρυξέλλες και θα μας πει ο κύριος Τίλεμαν στις απόψεις τους. Να πω επίσης ότι με χαρά διαπιστώσαμε ότι δύο τέος υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλαν επιστολές στην Lady Ashton για την σημασία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακούγεται με μια φωνή σε θέματα πανανθρωπίνων αξιών και δικαιωμάτων του ανθρώπου και ότι αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις δραστηριότητες της υπηρεσίας αυτής και στις σχέσεις της με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι επιστολές αυτές απεστάλησαν από τον κύριο Βέστερ Βέλε από πλευρά της Ομοσπονδιακής Γερμανίας και από την κυρία Έσπερσεν, την Υπουργό Εξωτερικών της Δανίας. Καλός για μια ακόμη φορά λοιπόν για να υπάρχει παρανόηση. Ο κύριος Βεστερβέλε είναι, ε, έκανα λάθος, δεν είναι ε, τέος υπουργό εξωτερικών της λαϊκής δημοκρατίας της Γερμανίας όπως προείπα, αλλά της Ομοσπονδιακής. Ο κύριος Τίλεμανς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. First and foremost, uh, I would like to point out uh, that δεν θα σας πω ότι είναι τιμή μου να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασίας στην ε, ε, Επιτροπή σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ε, ένα θεσμικό όργανο το οποίο ενδιαφέρεται πάρα πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε γι' αυτό το λόγο θέλουμε να δούμε πώ θα προβάλλουμε τη δράση των ανθρώπινα δικαιώματα και να δούμε τι θα γίνει και με την απονομή του Βεβίου Ζαχαρόφη για την ελευθερία της σκέψης, γιατί είναι κάτι το οποίο προσωπικά με έχει απασχολήσει. Είναι θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Γι' αυτό και έχουμε προσπαθήσει παντού να ε, προωθήσουμε την υπόσταση των ορμήνων για όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επομένως θα πρέπει να υπάρξει υποπτία, θα πρέπει να έχουμε για την επόμενη εξάμεινο συνεργασία να ανταλλάξουμε συμβουλές ε, και υπολογίζουμε πάρα πολύ στη βοήθεια της Επιτροπής σας. Να σας πω τι γίνεται όσον αφορά το έργο της ε, ψηλής εκπροσώπου όπως και εσείς αναφέρατε και έχουμε αυτή την ε, προσέγγιση που είναι μια κοινή προσπάθεια του Βελγίου και της υπηρεσίας της κυρίας Άστον. Βεβαίω και θα πρέπει να καλύψουμε, να λάβουμε υπόψη το τι έχει κάνει η Ισπανική Προεδρία και πρόκειται το Βέλγιο να καλύψει ε, αυτή την ε, πτυχή του έργου της κυρίας Θα ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο νωρίς και όσον αφορά τα πιο πρακτικά θέματα έχουμε γραμματεία από Βέλγιο, από Συμβούλιο και από Επιτροπή, οπότε θα δρούμε στις Βρυξέλλες, στην Γενέβη και στην Νέα Υόρκη. Με μεγάλη μας χαρά θα μας επικουρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτό πάντοτε είναι καλό σημάδι για μας ούτω ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το τόσο αξιόλογο έργο Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπόνηση του προγράμματος. Επίσης πρέπει να σας τονίσω ότι παντού η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία τώρα ε, έχει αναλάβει να προωθήσει το έργο μας. Έχουμε σε 10 χώρες ε, αντιπροσωπείες εμείς σαν Βέλγιο και έτσι κυρίως θα γίνουν μέσω αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι Βελγίου. Ε, δυνάμει της συνήθειας Λισαβόνας οι διαβουλευσει οι επαφές με τις τρίτες χώρες και με τους περιφερειακούς οργανισμούς πρόκειται να γίνονται με κυρίαρχο ρόλο των υπηρεσιών της κυρίας Άστον. Το ΔΕ Βέλγιο θα συμμετάσχει σε αυτές τις συναντήσεις σαν α, προεδρία της ΚΟΧΟΜ. Εδώ έχουμε μια σημαντική αλλαγή. Κατά το δεύτερο εξάμεινο ΔΕ του 2010 θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε και να παγιώνουμε την άσκηση αυτής της πολιτικής ανθρώπινων δικαιώματα της Ένωσης και θα δούμε πώς θα υπάρχει εφαρμογή αποτελεσματική των όσων σήμερα προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που δίνει η Συνθήκη της Λισαβόνας για να αυξήσουμε τις προσπάθειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις ε, αξίες τις οποίες πιστεύουμε στην εξωτερική πολιτική. Η αντιπρόεδρος, στις 16 έκτου στο Στρασβούργο ενώπιόν σας ε, δήλωσε ότι ενδιαφέρεται πρώτα όταν κάνει μία, έναν ε, απολογισμό της ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας είπε πώς θα μπορέσει να γίνει μία εκβάθρον αναθεώρηση και με την ευκαιρία να υπάρξουν καινούργιες καθημερινές γραμμές συνολική αναθεώρηση επομένως στα πλαίσια της COHOM. Ε, και έτσι θα έχουμε έργο προπαρασκευαστικό για τις ε, αποφάσεις τις οι οποίες θα ακολουθήσουν για να επιφέρει κάποιες αλλαγές. Βεβαίως, και το πρόγραμμα εργασίας δεν ε, λάβουμε υπόψη μόνο αυτού του τις επιτυχίες, αλλά και αυτή την επιστολή που αναφέρατε που περιέχει μια σειρά από ενδιαφέρουσες προτάσεις. Θα το χρησιμοποιήσουμε σαν βάση για τη συνέχεια. Σε αυτή την αναθεώρηση επίσης θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με όλους τους ε, εμπλεκομένους. Επίσης να δούμε τι θα γίνει με αυτό το ετήσιο φόρουμ των μη κυβερνητικών οργανώσεων στις 12 και 13 Ιουλίου, είναι στο τους. Ονομάζεται αυτό το φόρουμ η Συνήθεια Λισαβόνα και τα μέσα πολιτικής για ανθρώπινα δικαιώματα, η κατάσταση των πραγμάτων και το μέλλον. Και για άλλη μια φορά σας καλώ να συμμετάσχετε, θεωρούμε ότι είστε ε, από τους ομιλητές κλειδιά σε αυτή την εκδήλωση. για το έργο μας. Νομίζουμε ότι η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών θα είναι ένα πάρα πολύ βασικό σημείο. Κάποιες συστάσεις, ε, κάποια κριτήρια της Διεθνούς Αμνηστίας όσον αφορά την αναθεώρηση για αυτό το, το ε, σύνολο των μέσων πολιτικής που θα έχουμε. Είναι κάτι που θα διαπνέει όλο μας το έργο. Και βέβαια θέλουμε να εμπλέγουμε την κοινωνία των πολιτών. Ήδη έχουμε συνάντηση διαβούλευση στις 7 Εβδόμου στην πρώτη 19 ε, και 20 Ιουλίου και έτσι θα ανοιχτούμε στην κοινωνία των πολιτών. address... Με τις ε, θεσμικές αυτές αλλαγές μπορούμε τώρα την ευκαιρία να προχωρήσουμε τη δουλειά μας όπως σας προανέφερα σε μια προηγούμενη συνάντηση. Έχουμε τέσσερι άξονε, Πρώτα απ' όλα την προσαρμογή τη μεθοδολογία, τη ΚΟΧΟΜ. Δεύτερον, εφαρμογή των μέσων ε, πολιτική, τη Ευρωπαϊκής σε όλε τι πολιτικέ, Τρίτον, να προαχθεί ο ρόλο Ένωση στην, ε, στον ΟΗΕ και τέταρτον τα ανθρωπινά δικαιώματα να μπουν σε όλες τις πολιτικές και να υπάρχει μια συνέπεια μεταξύ ε, πολιτικής και ανθρωπινά δικαιώματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εσωτερική και εξωτερική πολιτική και γενικά στην ασκούμενη πολιτική και σε πιο συγκεκριμένες ε, εκφάνσεις της. Τώρα, ε, επιτρέψτε να μπω λίγο στις λεπτομέρειες. Για την ΚΟΧΟΜ πρώτα θα έχουμε περισσότερες ε, συναντήσεις, θα αυξάνεται η δουλειά και η ένταση του έργου του Συμβουλίου από τις Βεξέλλες, με τα κράτη-μέλη, ελπίζουμε να υπάρχει συνένεση για όλα αυτά, αλλά πάντως για πρακτικούς καθαρά λόγους μόλις καταρτιστεί το πρόγραμμα εργασίας θα δείτε ότι θα έχουμε συναντήσεις πιο συχνές. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μα και θα δείτε ότι αρκά και γρήγορα πρόκειται να πάρουν τα πρώτο δρόμο του επίση για την προσαρμογή τη μεθοδολογία, θα δούμε τι θα γίνει το σύστημα των Task Force, πώ θα έχουμε επιχειρησιακή λειτουργία, πώ θα προβάλλουμε την στρατηγία μα προ τα έξω, πώ θα μπορέσουμε να έχουμε ε, περισσότερη εμπλοκή τη Κορεπέρ τη επιτροπή Ασφάλειας και τελευταίο αλλά σημαντικό πώς θα μπορέσουμε έγκαιρα να αρχίσουμε τις επαφές για θέματα προτεραιότητας σε επίπεδο διπλωματικό. Ε, δεύτερον, όσον αφορά τα μέσα πολιτικής Ένωση, έχουμε δύο επιμέρου ζητήματα. Εξορθολογισμό και ένταξη αυτών των καθημερινών γραμμών σε όλες τι πολιτικέ. Δεύτερον, αναφέρει στο διαλόγο για των ε, διαβουλεύσεων. Σας είπα για τις επαφές με τη ΣΥΠΑ, κάτι το οποίο θα καλύψουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι αυτές τις πρακτικές που θα πρέπει να μπουν στο παιχνίδι και έχουμε αυτές τις καθητήριες γραμμές, την αναθεώρηση, την προσπάθεια ε, για ε, βελτίωση απόδοσής μας αλλά δεν καλύπτεται εδώ η αντιμετώπιση των κρίσεων των ένοπλων συγκρούσεων και ηχείως για το ρόλο των ανηλίκων σε αυτές τις ε, συγκρούσεις για την θανατική ποινή οπότε και πρόκειται να προωθήσουμε ψήφισμα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και εκεί θεωρούμε ότι θα τα πάμε καλύτερα σε σχέση με το 2007, τότε που για πρώτη φορά υπήρξε τέτοιο ψήφισμα. Και έτσι πιστεύουμε ότι πάρα πολλέ χώρε θα στηρίξουν ε, το, το, το, μορατόριο ε, σε σχέση με την ε, θανατική ποινή αλλά και στη συνέχεια προχωρήσουν για την κατάργηση. Η Ισπανική Προεδρία έκανε πάρα πάρα πολλά και σημαντικά για όλους τους τομείς που θέλουμε να ασχοληθούμε. Κοινωνία των πολιτών, οργανώσεις ενός δικαιώματα. Ε, όλοι αυτοί συνεννήθηκαν με τους εκπροσώπους της Ένωσης καθώς και την, είχαμε και την πρωτοβουλία εκείνη. και να δούμε και πώς θα μπορέσουμε να έχουμε το επιπλέον προεδρικό πρωτόκολλο όσον αφορά τα δικαιώματα των ενηλίκων γιατί θα υπάρξει και ένα δεύτερο πρωτόκολλο ούτω ώστε να έχουμε έναν μηχανισμό παραπώνων ο οποίος θα συγκροτηθεί. Επίσης να δούμε τι συνέχεια θα δοθεί και στα πρόσφατα συμπράσματα του Συμβουλίου. Επίση, να δούμε πώ οι καθημερινέ γραμμέ θα εφαρμοστούν και σε τοπικό επίπεδο. Αυτό που έχει ξεκινήσει η Σουηδική Προεδρία και θα έχουμε και την παρουσίαση τη Σουηδική Προεδρία. Αυτή η προσπάθεια κατά των βασανιστερίων. Βία τώρα κατά των γυναικών και διακρίσει, η ΚΟΧΟΜ και αυτό θα το εξετάσει και σε περιφερειακό επίπεδο. Εφαρμογή των καθημερινών γραμμών, ανταλλαγή πληροφοριών με τον νέο ειδικό εκπρόσωπο για τη σεξουαλική βία κατά τον Και η Επιτροπή επίσης είναι ένας άλλος τομέας που μας ε, απασχολεί, η δική σας υποεπιτροπή, αλλά έχουμε τους εξής έχουμε διαλόγους που επιτροπές, επαφές που θα γίνουν ε, την επόμενη, την επόμενη, διάρκεια. Ρωσία, ε, Λευκορωσία, Μολδαβία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία και Καζακστάν. Κουρδιστάν, Τατζικιστάν, Κίνα, με τη ΣΥΠΑ, με τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Χιλή, την Κολομβία, την Καμπότζη, το Λάος, το Βιετνάμ και το Μαρόκο. Και θέλω να επισημάνω πως η γραμματεία του Συμβουλίου θα κάνει αυτούς τους διαλόγους και θα συνεχίσουμε τη μελέτη του κινέζικου διαλόγου και του ρωσικού διαλόγου. Υπάρχουν και άλλα μέσα βεβαίως που πρέπει να αναφέρουμε για την ε, άνοιξη θρησκεία. Θα δούμε τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και θα συσταθεί μια προσωρινή ομάδα κρούσης για να εξετάσει το σχέδιο δράσης που προέκυψε από αυτά τα συμπεράσματα. Για την υποστήριξη της δημοκρατίας αναμένουμε έκθεση προόδου από τις υπηρεσίες της Αντιπροέδρου συμπεριλαμβανομένου ενό καταλόγου των χωρών αυτών στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας και ελπίζουμε να περάσουμε στην επιχειρησιακή φάση όσον αφορά τα ζητήματα ΛΟΑΤ χαρήκαμε που είδαμε ε, πώς μπορέσαμε να ευθύσουμε μια σειρά εργαλείων και βέβαια η προτεραιότητα μας θα είναι να εφαρμοστούν αυτά για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις για να υιοθετηθεί ένας κώδικας συμπεριφοράς ε, για τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα για να δρουν σύμφωνα με τη χάρτα τη σχετική του ΟΗΕ και ελπίζουμε να οριστικοποιηθεί και να εγκριθεί μέσα στους ερχόμενους έξι μήνες. Τρίτος τομέας προώθηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίπεδο του ΟΗΕ, οτιδήποτε σχετίζεται με τη Νέα Υόρκη και τη Γενέβη. Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γενική Συνέλευση. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι τη αναθεώρηση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σκοπεύαμε βεβαίως να ξεκινήσουμε το 2011, αλλά η εφετηρία θα είναι τότε. Η Ισπανική Προεδρία ήδη έχει δουλέψει πολύ εκεί. Οπότε πρέπει να δούμε την ρεαλιστική αλλά φιλόδοξη, το φιλόδοξο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτος τομέας και τελευταίος ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνοχή εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής θα ήθελα να αναφέρω πάλι κάποια ζητήματα προτεραιότητας. Πρώτα απ' όλα πώς να ενσωματωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΚΕΠΑ. Δεύτερον, γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια. Τρίτον, ελευθερία έκφρασης και νέες τεχνολογίες. Τέταρτον, ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρήσεις. Πέμπτον, δικαίωμα στο φαγητό σε όλους αυτούς τους τομείς. Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες τώρα, αλλά έχουμε σαφείς στόχους και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και βεβαίω είμαι και στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Τέλος. Τέλος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που δώσατε στην Κοχόμ τη δυνατότητα είναι το πρόγραμμα εργασίας, έχει ήδη διανεμηθεί. Το ελέγχουν σε αυτή τη φάση τα κράτη-μέλη και για μια ακόμη φορά σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αυτού του φιλόδοξου αλλά ρεαλιστικού προγράμματος θα έρθουμε σε επαφή και με την κοινωνία των πολιτών. Νομίζω είναι καλή η συγκυρία, λέει η Πρόεδρος. Με χαρά ακούσαμε ότι έχετε μια στρατηγική αντίληψη για την κατάσταση. Φυσικά και η Ισπανική Προεδρία έκανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και ευχαριστούμε τον κύριο Ντουάρτε ιδιαίτερα. Αλλά έχουμε την δυνατότητα να λειτουργήσουμε σε στρατηγικό επίπεδο πλέον. Αναφερθήκατε στα θέματα της στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την εφαρμογή και το streamlining των υπαρχών των μέσων Ελπίζω να συνεργαστούμε στενά στο μέλλον και θα είχα και μια ιδέα την οποία θα ήθελα να σας προτείνω για αξιολόγηση καταρχάς. Ίσως να μπορέσουμε να οργανώσουμε ένα κλειστό, ένα κλειστό σεμινάριο γύρω από τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του πού μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Ίσως λοιπόν από κοινού να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε μαζί, μιας και εμείς εξετάζουμε με οριζόντιο τρόπο σε αυτή τη φάση το θέμα των διαλόγων. Υπάρχουν και άλλοι τομείς τους οποίους θέλουμε να προχωρήσουμε και εδώ θα πρέπει να δείτε γενικότερα το θέμα της συνεργασίας με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ε, το mainstreaming είναι κάτι το οποίο μας αφορά ιδιαίτερα. Έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας σε σχέση με το, το δικαίωμα στην τροφή και με την ε, ασφάλεια στα τρόφιμα. Και έχει και αυτός τις ίδιες αντιστοιχίες. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Διεθνούς Αμνηστίας να μας μεταφέρει τις απόψεις ε, της Διεθνούς Αμνηστίας ε, για ε, το πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο ακούσαμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι πράγματι το πρόγραμμα αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε, εκτιμούμε θετικά και στην επιστολή των τέος, ε, των τέος Γερμανού και Δανού Υπουργού. Ε, νομίζω ότι ακούσαμε πράγματα τα οποία μας ικανοποίησαν. Το ίδιο ισχύει και για τον προεδρεύοντα του ΚΟΧΟΜ. Έχει κάνει αρκετά ανοίγματα το ΚΟΧΟΜ στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και στη δική μου οργάνωση, τη Διεθνή Αμνηστία, αλλά και στα δίκτυα σε σχέση με την συνεργασία μας τους επόμενους έξι μήνες θα ήθελα να ζητήσω να υπάρξει μεγαλύτερη, η μεγαλύτερη γενική διαφάνεια σε σχέση με τα έγγραφα των οποίων την πρόσβαση χάσαμε τους τελευταίους μήνες. Δεν κατηγορούμε την Ισπανική Προεδρία γι' αυτό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά θεσμικά θέματα που τίθενται τους τελευταίους μήνες. Ελπίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να προσπαθήσουμε να βρεθούμε πάλι στη φάση στην οποία είχαμε βρεθεί κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας όπου είχαμε πρόσβαση σε εσωτερικά έγγραφα, υποστηρικτικά έγγραφα, μνημόνια και ε, πολλές φορές και σε πρακτικά συναντήσεων υπουργών και τώρα που εργάζεστε στην υπηρεσία της ε, εκπροσώπου για τα εξωτερικά θέματα νομίζω ότι θα μπορέσετε να ενημερώσετε καλύτερα και το Κοινοβούλιο και τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ δύο έγγραφα στα οποία αναφερθήκατε. Καταρχάς, πρώτα οι δικές μας συστάσεις για την Φελγική Προεδρία δεν ξέρω αν δεν έχει διανεμηθεί σε όλα τα μέλη, θα γίνει η διανομή σήμερα. Υπάρχει και ένα σετ συστάσεων από το δίκτυο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό προς την Βελγική Προεδρία. Ιδιαίτερα για την περιοχή την Ευρωμεσογειακή. Δεν θα περάσω τώρα σε όλες τις λεπτομέρειες δεν θα ήθελα να μπω επίσης και σε θέματα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ξέρω ότι θα ακολουθήσει συζήτηση αργότερα γύρω από αυτό. Δεν θα ήθελα να ασχοληθούμε με θέματα κάπως πιο δύσκολα. Α, πάντως ξεκινώντας για την αναδιάρθρωση της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ανακοίνωσε η Lady Άστον πριν από δύο εβδομάδες, αυτό είναι κάτι που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ταιριάζει με την έννοια της αναθεώρησης την οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΚΟΧΟΜ. Και με το φόρουμ επίσης το οποίο θα οργανώσουμε εμείς τις επόμενες εβδομάδες. Ελπίζω λοιπόν να τεθεί σοβαρότατα και το θέμα των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που τέθηκε και από τον πρόεδρο του ΚΟΧΟΜ και από την πρόεδρο της Υποεπιτροπής. Υπάρχει πληθώρα διαδικασιών διαλόγου. Κάποιες από αυτές τις διαδικασίες είναι θετικές, είναι καρποφόρες που εφαρμόζονται από την τρίτη χώρα με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες άλλες διαδικασίες είναι απλά διπλωματικές προσπάθειες, διακοσμητικές ουσιαστικά. Δεν σημαίνει βέβαια δεν έχουν κανένα ρόλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν άλοθη για να μην υπάρχουν άλλες πολιτικές. Ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια μιας ευρύτερης αντίληψης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε συγκεκριμένες περιοχές Πάρα πολύ συχνά σε αυτή τη φάση έτσι αντιμετωπίζεται δυστυχώς ιδιαίτερα από τα κράτη-μέλη. Ένα βασικό θέμα είναι επίσης και η εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών, η καλύτερη εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών. Αυτό είναι κάτι που οι, κυβε... οι οργανώσεις, οι μη κυβερνητικέ ζητάνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι θα βγει τώρα από όλα αυτά ίσως μια μεγαλύτερη υπογράμμιση της σημασίας των τοπικών και ε, περιφερειακών στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει οι στρατηγικές αυτές να καλύψουν ε, τις τοπικές ανάγκες, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας με πιο ολοκληρωμένο τρόπο από ό,τι αυτόν που χρησιμοποιούμε σήμερα. Θα είναι ενδιαφέρον να δει κανείς πώς η κοινωνία των πολιτών μπορεί να ε, οργανώνει διαβουλεύσεις που να ενάσσονται σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Και αυτό η πρώτη απόδειξη θα είναι το Φόρουμ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 3ης Ιουλίου και θα υπάρξουν μάλιστα και δύο ε, ομάδες εργασίας που θα συνεδριάσουν. Η μία φορά την εσωτερική και εξωτερική συνοχή στα λαμβανόμενα μέτρα. Αυτό είναι κάτι που σαν Διεθνής Αμνηστία ζητάμε να υπάρξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και είναι θετικό να βλέπει κανείς ότι σαν θέμα ε, να γνωρίζεται το θέμα της συνεκτικότητας των διαδικασιών που ακολουθούνται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βγούμε από την ομάδα αυτής εργασίας με αρκετές ιδέες χρήσιμες. Μια άλλη ομάδα εργασίας πολύ ενδιαφέρουσα είναι αυτή που ασχολείται με το SCR. Ξέρω ότι αυτά τα θέματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα για τα θεσμικά όργανα επίσης και για μας στην Διεθνή Αμνησία ασχοληθήκαμε με αυτά μόνο τα τελευταία χρόνια ε, σε βάθος. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει συνολικά τα ανθρώπινα δικαιώματα από εδώ και πέρα, ε, δείχνοντας ότι είναι καθολικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην συγκεντρώνει την προσοχή της μόνο στα πολιτικά δικαιώματα όπως έκανε στο παρελθόν παραβλέποντας τα υπόλοιπα. Τώρα για τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου έχουν υπάρξει προβλήματα και στη Νέα Υόρκη αλλά κυρίως στη Γενέβη. Ελπίζουμε τα προβλήματα αυτά όχι μόνο σε επίπεδο αντιπροσωπευτικότητας αλλά και σε επίπεδο συντονισμού και σε επίπεδο υπολόγων ευθύνη για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί να ξεπεραστούν το ταχύτερο δυνατόν. Νομίζω ότι βασικό θέμα είναι το, ε, το Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Πάντα για τα Ηνωμένα Έθνη, κάτι το οποίο έχει υπογραμμιστεί βέβαια, είναι το ψήφισμα της ομάδας των 8 για τη θανατική ποινή. Ακούμε με μεγάλη χαρά ότι θα προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει προς την κατεύθυνση αυτή σαν βασική προτεραιότητά της. Έχουμε αρκετές ανησυχίες βέβαια ότι η διαδικασία δεν πηγαίνει με την ταχύτητα που θα έπρεπε θα ελπίζαμε να είχαμε προχωρήσει πολύ περισσότερο από ότι εκεί που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο, στο οποίο θα δραστηριοποιηθούμε εκ νέου και εμείς για συγκεκριμένες τρίτες χώρες. Νομίζουμε λοιπόν ότι μπορούμε να σημειώσουμε κάποια βήματα προόδου πριν από την Γενική Συνέλευση, γιατί αν περιμένουμε να δράσουμε μετά τη Γενική Συνέλευση, φοβάμαι ότι δεν θα, έχουμε κάνει τα βήματα που απαιτούνται. Κάποια επιπλέον σημεία. Ε, οι διμερείς συναντήσεις και επαφές. Λόγω όλων αυτών των θεσμικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο εξάμεινο, δεν έχουν υπάρξει πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις. Πολλές έχουν αναβληθεί. Το καταλαβαίνουμε αυτό, καταλαβαίνουμε το λόγο. Θα υπάρξουν ε, και υπήρξαν λίγες υπουργικές διμερείς συναντήσεις. Έχουμε βέβαια τη συνάντηση κορυφής για τη Μεσόγειο και ότι οι υπουργικές δομές τη συνοδεύουν. Όπως γνωρίζετε όλοι, πολλά από τα προβλήματά μας οφείλονται στο ότι πολλές από τις διμερείς υπουργικές συναντήσεις δεν οργανώνονται από την Κοχώμα αλλά από άλλες γεωγραφικές μονάδες. Και αυτό ε, είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει επιληθεί θυμίζω ακόμα και γι' αυτό εκτιμήσαμε αυτά τα οποία ο εκπρόσωπος της Κοχόμ και θα θέλαμε η παρουσία σας να χαρακτηρίζει πλέον και η μέθοδος εργασίας σας και αυτές τις συναντήσεις. Όπως συνέβη και με τις συστάσεις που δώσαμε προς την Ισπανική Προεδρία, περιλαμβάνουμε 10, στο τέλος 10 συγκεκριμένες περιπτώσεις. 10 συγκεκριμένες περιπτώσεις οι οποίες καλύπτουν θα έλεγα το σύνολο των ευρωπαϊκών μέσων και της ευρωπαϊκής εκδοχής με τρίτες χώρες και έχουν θα έλεγα καθολικό και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Περιμένουμε μηνύματα από τα θεσμικά όργανα σχετικά με την εφαρμογή και την χρήση όλων των μέσων αυτών στις 10 αυτές περιπτώσεις. Και περιμένουμε επίσης και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί συγκεκριμένα και να ζητήσει ενημέρωση για τις 10 μεμονωμένες αυτές περιπτώσεις τις οποίες έχουμε στο τέλος των συστάσεων. Ευχαριστώ, Ντέιβιντ. Πράγματι, όπως λες, η πρώτη ευκαιρία για να συναντηθεί η κοινωνία των πολιτών οικόχων και η υποεπιτροπή θα είναι 12 και 13 Ιουλίου στο φόρουμ των ΜΚΙΟ οπότε σε ευχαριστούμε θα έρθουμε πολύ από εμάς οπωσδήποτε τώρα λοιπόν να δώσω τον λόγο συναδέλφους κύριε Κάλκος βλέπω έχει ζητήσει το λόγο αλλά δεν είναι εδώ κάποιος άλλος Όχι. Κυρία Κιλ Νίλσεν. Ε, δεν είμαστε και πολλοί που θέλουμε το λόγο. Όσα ακούστηκαν είναι πολύ ενδιαφέροντα και σας ευχαριστώ. Δεν έχω ερωτήσεις να θέτω. Είμαι ικανοποιημένη από την παρουσίαση του Κοχών και θα ήθελα με αφορμή Αυτά να πω ότι η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε στείλει μια αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη για το μόνιμο φόρουμ των αυτοχθόνων. Θα πρέπει λοιπόν όταν μιλάμε για την αναθεώρηση και τις τροποποιήσεις στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα να μην ξεχνάμε ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν αυτόχθονες λαοί και εμείς σαν Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τίλεμανς θα ήθελε να αντιδράσει σε αυτά που ακούσαμε. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και ζήτημα πιο ενισχυμένη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι κρίμα που δεν το ανέφερα αυτό τη συνεργασία με την υποεπιτροπή σας δηλαδή στην αφορά μου. Σας προσκαλέσαμε και εμείς για μια συνεδρίαση της ε, ΚΟΧΟΜ που θα λάβει χώρα το φθινόπωρο για να συζητήσουμε τις ε, θεσμικές αλλαγές ε, που επέφερε η συνθήκη της Λισαβόνας στην σχέση των θεσμικών οργάνων. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ραντεβού αυτό για μας. ιδέα τώρα ενό σεμιναρίου και ενό εργαστηρίου είναι πολύ ενδιαφέρουσα. για να έχουμε και συνεννοήσεις με την κοινωνία των πολιτών. Γεγονός είναι πως οι διάλογοι είναι και οι διαβουλεύσεις είναι πολλές, αποτελέσματα κειμένονται και η αναθεώρηση που πρέπει να γίνει αφορά το πώς, πώς θα προχωρήσουμε αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα οτιδήποτε νέες ιδέες είναι ευπρόσδεκτες γιατί καμιά φορά υπάρχει η τάση έτσι κάπως συντηρητικοί όσον αφορά τους διαλόγους. Και για όλη διαδικασία χρειάζεται κάποια συνεισφορά εξωτερική εξωτερική δεσπάνω σε σχέση με την παραδοσιακή λειτουργία και βεβαίως για το διάλογο και τη διαβούλευση θα ακούσουμε και τα σχόλια της Κομισιόν σημειώνω αυτά τα οποία είπε η Διεθνή Αμνηστία. Ίσως είναι ζήτημα διαφάνειας. τόσο αν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αστείευτηκα. Αλλά είναι έξυπνο αυτό. Γιατί τι επισημαίνουμε. Όπως είδε και ο David τους τελευταίους έξι μήνες οι oh. μετασχηματισμοί αυτοί προκαλούν και ανοργανωσιά and I do not expect that in the following six months will uh, bring full clarity. Και δεν περιμένω έτσι, τους επόμενους έξι μήνες να έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ε, ακόμα οργανωνόμαστε. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε και επειδή είναι και το κοινό Κοινοβούλιο ένα σοβαρό θεσμικό όργανο και η κοινωνία των πολιτών βεβαίω ε, θα μας απασχολήσει θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γνωρίζοντας πως υπάρχει χρειάζεται βεβαίω ε, μια διαδικασία προσαρμογής Τώρα, για τη θανατική ποινή είχαμε μια καλή πρώτη συνάντηση της σχετικής ομάδας στη Νέα Υόρκη και τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής συνάντησης μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Να επισημάνω επίσης πως στη Γενέβη και στη Νέα Υόρκη είχαμε ξεκινήσει να εργαζόμαστε αλλά να σας πω πως ε, η αντιπροσωπεία της Ένωσης ε, είναι συνεννόηση με τη βελγική αντιπροσωπεία ο σχεδιασμός, προγραμματισμός άλλο ένα βήμα λοιπόν προς την υπηρεσία εξωτερικής δράσης Αυτά λοιπόν νομίζω πως αρκετά μίλησα. Ευχαριστώ. Uh, Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Γκέρενς και μετά στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν θέλουν συνάδελφοι μπορεί να επανέλθουν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έφτασα με καθυστέρηση και δεν ξέρω αν είχατε την δυνατότητα να συζητήσετε το θέμα της ένταξης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα κεφαλαιόδες για όλους μας και αυτό για πολλούς λόγους. Πρώτον, πρόκειται για μια δήλωση πίστης, αν θέλετε, των 27 σε κοινέ αξίες. Πόσο μάλλον που αυτό γίνεται στα πλαίσια των εξωτερικών μας σχέσεων. Νομίζω ότι μπορέσουμε να δράσουμε ομαδικά και να πετύχουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να πετύχουμε στο παρελθόν. Θα πρέπει βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς αυτό να είναι, ε, θα έλεγα, αξιόπιστη. Εμένω σε ένα θέμα, εδώ και πάρα πολύ καιρό και γίνομαι κουραστικός, το καθήκον για όλες τις χώρες να δεχθούν όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε στους Ρώσους στα πλαίσια των εξωτερικών μας σχέσεων και των σχέσεων καλής γειτονίας ή στα πλαίσια μιας συνάντησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας ότι θα πρέπει να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ κάποιες από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι διατεθειμένες να δεχθούν τις αποφάσεις του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Υπάρχει εδώ μια αντίφαση. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η Βελγική Προεδρία έτσι ώστε να, να έλεγα να αλλάξει αυτός ο αναχρονισμός. Μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες και να υποχρεώσουμε τους 27 να σεβαστούν όλες τις αποφάσεις για του, του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Επιμένω σε αυτό και επιμένω σε αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Κύριε Γκέρενς, νομίζω ότι καλά κάνετε και επιμένετε. Είναι χρήσιμο που επαναλαμβάνετε αυτά τα πράγματα και σαν πολιτικός ξέρω ότι κάποιοι πρέπει να επαναλαμβάνουν ορισμένα θέματα και τότε μόνο θα τα δουν να πραγματοποιούνται. Νομίζω είναι καλή ιδέα να εκφράσουμε μια κάποια επιθυμία μας σε σχέση συγκεκριμένη επιθυμία μας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή ε, Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν τα είχαμε συζητήσει πρόσφατα αυτά τα θέματα. Λοιπόν κύριε Τίλεμαν, έχετε χρόνο να σκεφτείτε την πρόταση Γκέρενς αλλά να ακούσουμε τώρα και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε our Belgian friends about the team spirit. I mean, never been uh, so involved before a Λοιπόν, καλό είναι που έχουμε τώρα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα που είναι εδώ παρούσα και τους γειτονές μας της ΚΟΧΟΜ. Λοιπόν, Νομίζω ότι η επαφή την οποία είχαμε με την Κοχόμ για τον καθαρισμό του προγραμματισμού της ε, είναι κάτι το πάρα πολύ καλό. Η εξάμηνη αυτή διάρκεια θα ξεκινήσει πάρα πολύ θετικά προγράμματα. Ε, όλα αυτά τα οποία θα ξεκινήσουμε βέβαια δεν πρόκειται να τα ολοκληρώσουμε μέσα σε έξι μήνες. Μια και μιλάμε για μια νέα στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί οι παλαιότερη είναι πλέον πεπερασμένη, είχε ξεκινήσει θυμίζω το 2001. Έχουμε λοιπόν το φόρουμ για την κοινωνία των πολιτών και της ΜΚΟ και στο τέλος του εξαμήνου νομίζω ότι θα έχουμε κάποια πράγματα να πούμε. Θα ήθελα επίσης να αντιδράσω λίγο σε τρία σημεία. Καταρχάς για την συνεκτικότητα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τη δράση μας. Είναι σαφές ότι αυτή είναι μια προτεραιότητα η οποία γίνεται αισθητή από όλους τους εμπλεκομένους. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα, ε, την Προεδρία της ΚΟΧΟΜ και τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά κυρίως την εξωτερική πλευρά. Έχουμε πορεία να, να διανύσουμε συγγνώμη, σε εσωτερικό επίπεδο έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλες τις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές του Κοινοβουλίου. Υπάρχει πολλή δουλειά που μένει να γίνει ακόμα και χαίρομαι που η κυρία Ντοκεζέρ ε, δέχτηκε να προεδρεύσει ε, μια ομάδα εργασίας για την εσωτερική και εξωτερική συνεκτικότητα στο φόρουμ για τα ΜΚΟ. Έχουμε επίσης το εξαιρετικό παράδειγμα του κ. Χούχεντς για τα θέματα της ε, ένταξής μας ε, ε, στην Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τελικά για μας όταν ερχόμαστε σε επαφή με τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούμε να δεχτούμε αυτόματα τον μηχανισμό ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Γι' αυτό παρακαλώ προχωρήστε προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στις σχέσεις με τις υπόλοιπες χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης. Ένα σημαντικό στοιχείο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι στις εξωτερικές σχέσεις υπάρχουν κάποια όρια βέβαια, αλλά από την άλλη δεν θα περιοριστούμε εμείς και θα αναφερθούμε σε όλα τα θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσωτερικά έχουμε αυτό που λέμε στα γαλλικά competence d'attribution, δηλαδή ε, συγκεκριμένες αρμοδιότητες να ξεκινήσουν σαν παράδειγμα συζητήσεις με διάφορες χώρες για την καθυστέρηση μεταφοράς της κοινοτική νομοθεσίας στην εσωτερική τους νομοθεσία. Έχουμε αυτές τις δυνατότητες κατανομής των προτεραιοτήτων. Έχουμε τις δυνατότητες για να ευαισθητοποιήσουμε αν θέλετε σε επίπεδο εσωτερικό. Αλλά έχουμε περιορισμούς ως προς το εξωτερικό και έχουμε και περιορισμού από την ίδια τη συνθήκη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο φόρουμ για τη ΜΚΟ. Ε, για τον διάλογο, ε, για τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένας αριθμός διαλόγων πάει καλά, ε, κάποιοι άλλοι διάλογοι δεν είναι παραπλές διπλωματικές ασκήσεις και υπάρχουν και μορφές διαλόγου οι οποίες θα έλεγα θεωρητικά θα μπορούσαν να είναι ουσιαστικό τμήμα των συμφωνιών για εταιρικές σχέσεις κτλ. Ε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το τι γίνεται σε σχέση με αυτό το κομμάτι για άλλα θέματα όπως οι εμπορικές σχέσεις. Ένα τελευταίο σημείο αφορά ε, τις εργασίες του Κοχόμ σχετικά με το πόσες φορές θα συνεδριάζει, που θα είναι η έδρα του κτλ. Είναι απαραίτητο νομίζω, ιδιαίτερα για το εξάμεινο αυτό, ε, διατρέχει ένα κίνδυνο η κατάσταση. Στην ουσία να χάσουν κατά κάποιο τρόπο την καθοδηγητική αν θέλετε αρμοδιότητα την οποία έχουν τα κράτη-μέλη σε σχέση με την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυρία Άστον για να μειωθεί έτσι, αυτό το φαινόμενο. Οπότε θα πρέπει να ακούσουμε τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουμε αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Κέρτς. Νομίζω πως ε, υπάρχει το ζήτημα που έθεσε ο Συνάδελφου είναι δύσκολο να έχουμε εμεί πρόσβαση στις δομές ε, και στι ομάδες εργασίας ε, του Συμβουλίου. Αυτό δεν εννοούσε, Ντέιβιντ. Πως ανθρώπινα δικαιώματα φαίνεται πως απουσιάζουν αυτό τι γίνεται στο Συμβούλιο και πρέπει να το φροντίσουμε τώρα που στείνεται η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Παρά το ότι θέλει βεβαίως να τα συνδέσει όλα αυτά η κυρία Άστον, φοβάμαι πως οι άνθρωποι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλοι με άλλα. Δεν είναι ιδανικό αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από σας Επίσης φοβάμαι πω ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Μακμίλαν Σκοτ, έφυγε ενώ ήμουν έτοιμη να ρωτήσω κάτι. Και αυτό αφορά την προώθηση της δημοκρατίας. Ξέρω πως εκπροσωπεί το κοινοβούλιο με τον πρόεδρο Μπούζεκ αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον σε ένα διάλογο υψηλού επίπεδου για την προώθηση της δημοκρατίας Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ρωτήσω τους κυρίους Τίλεμανς και Χέρτς εάν ασχολούνται με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη στήριξη της ε, Δημοκρατίας. Δύο πράγματα, λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω και μετά στις 10.30 θα ξεκινήσει η ακρόαση για το Κονγκό. Ο κύριος Τίλεμανς. Να αναφερθώ λοιπόν στα ερωτήματα του κυρίου Βουλευτού. Μα γι' αυτό ασχολούμαστε με το ζήτημα της εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μας δίνει πρώτα απ' όλα τη δυνατότητα να υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ΕΣΔΑ και τη χάρτα και η χάρτα βεβαίως της Ένωσης ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει τεθεί ενισχύ πλην των χωρών εκείνων που έχουν opt-out. Ε, τα δύο αυτά ζητήματα Εμείς θα συζητάμε όσον αφορά την συνοχή της πολιτικής και βέβαια θα δούμε και τις επιτροπές που επιτερώνουν συνθήκες του ΟΗΕ. Και θα θέσω το ζήτημα με την άδειά σας έτσι ώστε η συμπεριφορά των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των συνθήκων του ΟΗΕ να ληφθεί υπόψη. Ένα τελευταίο σημείο. Το ΚΟΕΣ, η ομάδα εργασίας δηλαδή που ασχολείται με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ, τα έχει εκεί φροντίσει αυτά. Τότε καλό είναι να έρθετε σε επαφή μαζί τους ε, για τις δύο γεωγραφικές ομάδες. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα όταν μιλάμε για έλλειψη διαφάνειας. Αυτό εννοούμε, αυτές τις ομάδες. Πρόθεσή μας είναι να ενσωματώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα περαιτέρω στις γεωγραφικές ομάδες. Πώς θα γίνει αυτό. Θα προσεγγίσουμε τους Βέλγους Προέδρους των ομάδων εργασίας και θα δούμε αν μπορεί η κοινωνία των πολιτών να τους μιλήσει άμεσα βεβαίως όλοι οι διάλογοι και οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να είναι να γίνονται από κοινού από την Επιτροπή και τις γεωγραφικές ομάδες και ελπίζουμε να έχουμε συζήτηση λοιπόν μεταξύ της ΚΟΧΟΜ και των γεωγραφικών αυτών ομάδων επίσης και τα θέματα προσπαθούμε να ενσωματώσουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα το δικαίωμα στο φαγητό. Προσπαθούμε π.χ. να συνεχίσουμε την Κοντεφ. Κοντεφ. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα συνεργασίας ε, με το Συμβούλιο. Ανθρώπινα δικαιώματα στην ΚΕΠΑ. Ένα άλλο παράδειγμα συνεργασίας με την ομάδα εργασίας. Ε, επίσης η ΣΥΡΚΟΜ ε, που είναι στην αρμοδιότητα της ε, Πολιτικής Επιτροπής και Πολιτικής Ασφαλείας και με αυτούς θα συνεργαστούμε στενά. Για τη δημοκρατία, η στήριξη της δημοκρατίας μας απασχολεί επίσης πάρα πολύ. Τι άλλο έχω να σας πω Διακόπτει ο μιλητής. So, Όπως είπα προηγουμένως, θα περιμένουμε και την έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εκπροσώπων του Συμβουλίου για τις λεγόμενες χώρες πιλότους. Οπότε το ζήτημα είναι να δούμε τα, τα συμπεράσματα και δεν ξέρω ίσως η Κομισιόν θέλει εδώ να πάρει το λόγο για αυτό το θέμα για το πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε συνέχεια στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για αυτό το θέμα και οπωσδήποτε κυρία Πρόεδρε θα σας ενημερώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τίλεμαντς, ο κύριος Σέρτς θέλει να πάρει το λόγο. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω για τη δημοκρατία. Πρέπει να κάνουμε μια έκθεση προς το Συμβούλιο και η ΚΟΧΟΜ θα τη λάβει νομίζω το Νοέμβριο και οπωσδήποτε θα συμπεριλάβουμε και το Κοινοβούλιο γιατί σας εκτιμούμε πάρα πολύ. Α, ε, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν αυτήν την ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Τίλεμανς και πρέπει να μάθω τον τίτλο σας γιατί είναι εντελώς νέος για μας. Πρόεδρος της ΚΟΧΟΜ στην υπηρεσία της ΥΠΑ του εκπροσώπου για την εξωτερική δράση. Uh, και υπεύθυνο για επαφές και με την κοινωνία των πολιτών και της ΜΚΟ. Μαζί νομίζω θα πετύχουμε πολλά. Συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο κύριο θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Είναι η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην δημοκρατία του Κονγκό αυτή την ακρόαση την οργανώνουμε σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανάπτυξης και καλωσορίζω την Πρόεδρό της εδώ. Γιατί είναι επίκαιρη η συνάντηση αυτή. Γιατί έχουμε να κάνουμε με τα 50 χρόνια της ίδρυσης της Δημοκρατίας του Κονγκό που γιορτάστηκαν χθες. 30 Ιουνίου. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και το κατεπήγον ψήφισμα που υιοθέτησε τον προηγούμενο μήνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά το φόνο του κυρίου Τσεμπέια. Αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση προκάλεσε την προσοχή όλων. Ήταν πράγματι ένας προασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέχρι την τελευταία στιγμή στη ζωή του ήταν ένας δικηγόρος ο οποίος δεν φοβόταν να ασχοληθεί με θέματα τα οποία ήταν ε, εναντίον των συμφερόντων αυτών που έχουν την εξουσία και πλήρωσε την προσπάθειά του με τη ζωή του. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο πρέπει να κάνουμε τη συνάντηση αυτή σήμερα είναι ότι η επόμενη συνάντηση ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινοβουλευτική, θα διεξαχθεί στην Κινσάσα στο Κονγκό από τις 2 μέχρι 5 Δεκεμβρίου του 2010. Τον προηγούμενο Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα κατεπήγων, γενικότερο θα έλεγα, Επίσης και το Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ έκανε την περιοδική έκθεσή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κονγκό τον Μάρτιο. Πολλές συστάσεις έγιναν δεκτές από την κυβέρνηση του Κονγκό και θα βρείτε την έκθεση στο φάκελό σας. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι ο ειδικό ε, εισηγητής για τις εξοδικαστικές εκτελέσεις των Ηνωμένων Εθνών ο κ. επισκέφθηκε τη Δημοκρατία του Κονγκό και δημοσίευσε τη δική του έκθεση η οποία αναφέρεται σε πολύ σημαντικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξοδικαστικές εκτελέσεις, δολοφονίες γενικότερα. Από το Δεκέμβριο του 2007 μέχρι το Μάρτιο του 2010, 1796 άμαχοι σκοτώθηκαν και 1777 έπεσαν θύματα απαγωγής από τους οποίους οι 700 περίπου ήσαν ανήλικοι. Υπάρχει ατιμορρησία, ε, οι αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις καταστολής ασκούν βία, υπάρχει επίσης σεξουαλική βία, ο βιασμός χρησιμοποιείται σαν μέσο διεξαγωγής πολέμου, 160 γυναίκες την εβδομάδα πέφτουν θύματα βιασμού, θύματα βιασμού και οι συνθήκες φυσικά φυλάκισης, κράτησης ε, είναι βασανιστικές και υπάρχει φυσικά και το θέμα των βασανιστήριων. Όλα αυτά μας οδηγούν στο να ε, εξετάσουμε την κατάσταση σε μια χώρα όπου υπάρχουν στο εσωτερικό της και σχεδόν δύο εκατομμύρια εκτοπισμένοι που προκαλούνται από την δράση ενόπλων ομάδων όπως ε, η ομάδα αντίστασης στο όνομα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόγραμμά μας. Εδώ έχω μαζί μου την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης και θα ήθελα να της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την οργάνωση αυτής της ακρόασης σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι και φιλοξενούμενοι, χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Συνεργασία. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κονγκό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Καλό είναι να συζητά κανείς τα βήματα προόδου που έχουν υπάρξει σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κονγκό, αλλά υπάρχουν όμως και πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με την κλιμάκωση της βίας στην περιοχή και αυτό μας απασχολεί. Έχουμε εξετάσει τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες αφορούν κυρίως την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και όπου δυστυχώς οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δυσκολεύουν πάρα πολύ την κατάσταση. Έχουμε καταδικάσει τα εγκλήματα τα οποία έχουν συμβεί στο Κονγκό και ζητάμε να υπάρξουν δημοκρατικές λύσεις για να τερματιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Έχουμε επίσης οργανώσει και μία ειδική συνάντηση για την κατάσταση των γυναικών στη Δημοκρατία του Κονγκό, γιατί οι βιασμοί εις βάρος παιδιών πολλές φορές, ε, κοριτσιών αλλά και αγοριών, και φυσικά γυναικών γίνονται σε καθημερινή βάση και είναι σε καθημερινή βάση η πραγματικότητα. Ο Επίτροπος Ντεγκούχτο, ο ε, αρμόδιος Επίτροπος, έχει ασχοληθεί και αυτός και έχει καταδικάζει τα απαράδεκτα αυτά φαινόμενα Έχουμε και την δολοφονία του συγκεκριμένου εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών, ο οποίος δεν έγινε αντικείμενο προστασίας από τα διεθνή δίκτυα προστασίας των πρωταγωνιστών για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όπως είπε η Πρόεδρος προστέθηκε το όνομά του στον ατελείωτο αυτό κατάλογο των θυμάτων φόνων δολοφονιών, εκτελέσεων και ε, ε, βιασμών. Κρίμα είναι που χθε είχαμε την 50η επέτειο από την ανεξαρτησία του Κονγκό και δεν έχει ποτέ υπάρξει ένα έτος δημοκρατίας. Υπάρχει μόνο φόβος για το αύριο. Επίσης δεν υπάρχει χρηματοδότηση και κινδυνεύουν έτσι οι ανθρωπιστικές ομάδες επιτόπου. Επίσης, εμείς πάντα αλλάζουμε προτεραιότητες, τέλος πάντων πρέπει να παραμείνει η δημοκρατία του Κογκό προτεραιότητάς μας. Αυτό σημαίνει δηλαδή πως οι δωρητές πρέπει να φροντίσουν το 70% από τα 825 εκατομμύρια δολάρια που έχει ζητήσει ο ΙΕ να δοθεί. Η δημοκρατία έχει χάσει πάρα πολλές μάχες στο Κονγκό Πρέπει λοιπόν όλοι να κάνουμε, πώς να γραμματίσουμε τη στρατηγική μας. κατά όλων αυτών των φαινομένων. Είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αρμοδίων επιτρόπων και της κυρίας Άστον να προωθήσουν αυτή τη στρατηγική για να βοηθήσουν τον ΟΗΕ. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κρετού. Τώρα θα προσκαλέσω τον πρώτο μας ομιλητή να μιλήσει για 10 λεπτάκια. Ο ομιλητής είναι ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρόεδρος της League des Electeurs του Κονγκό, ο κύριος Πόλ Ζαμοκούα έχετε τον λόγο. Και όσοι μπορείτε να δείτε τον κύριο Μούκουα, βλέπετε πως δίπλα του έχουμε τη φωτογραφία του κυρίου Τσεμπέγια. Mesdames et messieurs les parlementaires, Κυρίες και κύριοι, κοινοβουλευτική εξ ονόματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των μελών οργανώσεων στην Δημοκρατία του Κονγκό, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που μου επιτρέψατε να συμμετέχω σε αυτή τη σημαντική δραστηριότητα για τη χώρα μου. Θα ήθελα προκαταρκτικά να σας πω ότι την 1η Ιουνίου, τη νύχτα της 1ης Ιουνίου, δύο υπρασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της οργάνωσης ε, φωνές αυτών που δεν έχουν φωνή. Οι κύριοι Τσεμπέγια και κύριος Μπαζάνα δολοφονήθηκαν. Ο πρώτος δολοφονήθηκε αποδεδειγμένο και ο δεύτερος πλέον έχει, είναι αγνοούμενος και μάλιστα μέσα στα γραφεία της ε, ε, Εθνικής Αστυνομίας στην Κινσάσα πάρα πολλές ενδείξεις ε, νομίζω μας οδηγούν στο να κατανοήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην κορυφή της κρατικής υποδομής της χώρας μου. Θα ήθελα αγαπητοί βουλευτές να τηρήσουμε στην ύμη τους ενός λεπτού σιγής. Αυτό το πρόσφατο διπλό πολιτικό έγκλημα θα έλεγα μεγαλώνει τον κατάλογο των πολιτικών δολοφονιών μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο Πολύκαρπος Πογγί, ο Πασχάλης Καλμπογκουλού, ο Σέρζ Μαχές, ο Μπαβούβα Μουάμπα και ο Ντιντάτς Ναμουζωμά δολοφονήθηκαν και αυτοί και αυτά όλα δείχνουν την κατάσταση στα πλαίσια της οποίας οι αρχές δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Δυστυχώς οι δολοφονίες αυτές δεν εκπλήσουν πλέον κανένα. Οι οργανώσεις μας είχαν προειδοποιήσει εδώ και ένα χρόνο τη διεθνή κοινότητα για την τεράστια πίεση και απειλή που υφίσταντο οι οργανώσεις αυτές. Τέσσερα χρόνια μετά από τις ελπίδες που προκλήθηκαν στις εκλογές του 2006, η διεθνής κοινότητα είχε στηρίξει τις εκλογικές διαδικασίες, αλλά δυστυχώς τέσσερα χρόνια μετά η κατάσταση που περιγράφουν ε, οι οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι φρικτή και αυτό αφορά το σύνολο του εδάφους της Δημοκρατίας του Κόγκο. Η κατάσταση αυτή είναι πιο δραματική στα ανατολικά της χώρας. Σήμερα όλοι οι δείκτες είναι πλέον στο κόκκινο και σε όλους τους τομείς τα πολιτικά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά. Ενώ θα αρκούσε μια απλή ε, βούληση πολιτική από πλευράς ε, της ε, κυβέρνησης και όχι τεράστια οικονομικά μέσα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν ότι ε, το άλοθη της περίοδου της μετασυγκρουσιακής την οποία χρησιμοποιεί συστηματικά η κυβέρνηση δεν είναι παρά ένα άλοθη το οποίο κρύβει την αποτυχία της κυβέρνησης να προστατεύσει τη δημοκρατία όλες οι επιθυμίες για αλλαγές δημοκρατικές έχουν μπλοκαριστεί από την ίδια την κυβέρνηση. Υπάρχει πλήρης καταστολή των δραστηριοτήτων της αντιπολίτευσης, της δραστηριότητας των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της απλής λειτουργίας των αντιπολιτευομένων μέσων ενημέρωσης καμία δημοκρατική ελευθερία δεν γίνεται σεβαστή και κανένα δικαίωμα δεν έχει πλέον η πολιτική αντιπολίτευση. Οι ειρηνικές διαδηλώσεις απαγορεύονται και όταν υπάρχουν καταστέλλονται βία. Και ε, ταυτόχρονα η κοινωνία των πολιτών ταυτίζεται με την αντιπολίτευση και γίνεται ο αντικείμενο συστηματικής ενόχλησης και καταστολής ε, συλλαμβάνονται και δολοφονούνται οι εκπρόσωποι της μέσα σε μια πλήρη ατιμορρησία από πλευράς δικαστικών αρχών. Έχει ξεφύγει η κυβέρνηση αυτή και ενισχύεται από την κατάρρευση του κράτους δικαίου διότι η δικαιοσύνη πλέον ανήκει στην πολιτική και από την άλλη υπάρχει και μια προφανής επιθυμία των αρχών να διατηρούν πολλαπλές μορφές τήρησης τάξης χωρίς περιορισμούς στην χρήση ε, βασανιστήριων και άλλων πρακτικών. Τα εγκλήματα τα οποία είναι πάρα πολλά και τα οποία οφείλονται θα έλεγα στη δράση της κυβέρνησης. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διαβάσετε προσεκτικά την τελευταία έκθεση της Ομοσπονδίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί λόγω της τάσης της κυβέρνησης της Κινσάσα. Ε, δεν θα ήθελα να ε, σας καθυστερήσω πολύ και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να περάσω στις συστάσεις που ανήκουν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις συγκεκριμένες τελευταίες δηλοφονίες και ιδιαίτερα την δολοφονία του Φλωριμπέρ Τσεμπεγιά. Οι δεύτερες ε, συστάσεις αφορούν τον πολιτικό διάλογο ευρωπαϊκή Ένωσης και Δημοκρατίας του Κονγκό και η τρίτη κατηγορία συστάσεων ε, αφορά το θέμα της συνεργασίας. Σχετικά με τη δολοφονία του Φλωριμπέρ Σεμπεγιά, η Διεθνής αυτή Ομοσπονδία και ε, τα μέλη της στο Κονγκό σας παρακαλούν να πιέσετε την κυβέρνηση στην Κινσάσα για να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη διεθνής ε, επιτροπή έρευνας. Σας ζητάμε επίσης να συνεισφέρετε στην προστασία της οικογένειας και των συγγενών του Σεμπεγιά και όλων αυτών οι οποίοι απειλούνται λόγω της δραστηριότητάς τους. Σας ζητάμε να απαιτήσετε από την κυβέρνηση την Κινσάσα και από τις αντιπροσωπείες των χωρών σας και της Ένωσης στην Κινσάσα να οργανώσουν κατεπηγόντως μία συνάντηση ανάμεσα στους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κυβέρνηση έτσι ώστε να καθοριστεί σωστά ο μηχανισμός προστασίας αυτών που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ζητάμε επίσης να ζητήσετε από τις πρεσβείες και την αντιπροσωπεία να, σε, να συμμετέχουν, να είναι παρούσες στις δίκες εις βάρος αυτών που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ζητάμε επίσης να εφαρμόσετε με πιο αποτελεσματικό και συγκεκριμένο τρόπο τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία αυτών που προσπαθούν να εφαρμόσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί πέρα από τη δολοφονία του Σεμπέγια και του Μπανζάνα, ο στόχος αυτών που μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι να μπορέσουν να λειτουργήσουν ελεύθερα. Είχε σταλεί μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινωνίας των πολιτών που είχε πάει στην Κινσάσα που διαπίστωσε την αποτυχία τελικά της προσπάθειας που έκαναν οι διεθνείς οργανώσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα πλαίσιο που θα επέτρεπε να λειτουργήσουν οι δομές για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ζητάμε επίσης και ικανομικά να βοηθήσετε τις ανεξάρτητες οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που από το 2006 δεν παίρνουν καμία χρηματοδότηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις συστάσεις για τον πολιτικό διάλογο με την δημοκρατία του Κονγκό. Θα ήθελα να σας προτείνω δύο βασικές συστάσεις. Πρώτον, να προχωρήσετε στην δημιουργία ενός πολιτικού διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας του Κονγκό, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συμφωνίας του Κοτονού που επιτρέπει να τεθεί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο κέντρο των σχέσεων των διπλωματικών ανάμεσα στην Ένωση και το Κονγκό και αυτό να γίνει με διαφανή αλλά επίσημο τρόπο σε συνεργασία και με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και τέλος να εμπλέξετε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην διαδικασία προπαρασκευής και συμμετοχής στον πολιτικό διάλογο σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συμφωνίας του Κοτονού. Θα ήθελα <coughs> να καταλήξω με δύο συστάσεις σχετικές με τις μορφές συνεργασίας. Θα ήθελα να σας ζητήσω καταρχάς να εμπλέξετε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και στην εφαρμογή των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Κονγκό, όπως το ΕΠΟΛ και το Ρετζίσκο. Θα θέλαμε επίσης να σας ζητήσουμε να εισάγετε συγκεκριμένα κριτήρια σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα προγράμματα συνεργασίας που διαπραγματεύεστε με τις αρχές του Κονγκό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορέσει και μέσω του δημοσιονομικού ελέγχου ότι τα χρήματα που δίδονται στις αρχές του Κονγκό συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην βελτίωση της κατάστασης στα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι στην ενίσχυση ενός δικαστικού συστήματος που χρησιμοποιείται σαν μέσο καταστολής εις βάρος των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενός συστήματος στήρησης τάξης που δεν είναι παρά μια μόνιμη πηγή παραβιάσεων της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Επιτρέψτε μου λοιπόν κλείνοντας κυρίες και κύριοι να σας ζητήσω να λάβετε υπόψη σας σοβαρά τις συστάσεις αυτές και όλες αυτές τις συστάσεις που περιλαμβάνονται τον τελευταίο καιρό στις εκθέσεις μας. Τότε μόνο θα μπορέσετε πραγματικά να συνεισφέρετε στην αμονομή δικαιοσύνης για την δολοφονία του Φλωριμπέρ Σεμπεγιά και την εξαφάνιση του Φιντέλ Μπανζανά και να βοηθήσετε έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ελεύθερες εκλογές στο Κονγκό. Στο όνομα λοιπόν της οργάνωσής μου και των εταίρων της σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να εκφραστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε, ο κύριος Λετέρν, ο πρώην Πρωθυπουργός, ζήτησε να υπάρχει κάποια τέτοια αντικειμενική ε, διερεύνηση της διεθνούς κοινότητας για τις δολοφονίες. Και αυτό και με την ευκαιρία της 50ης επαιτίου της εξαρτησίας της χώρας. Και τώρα έχουμε τον απεσταλμένο του κυρίου του, του, του, του, κύριε Γκότσαλκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Ονομάζομαι Γκόσολτ. Μιλάει πάρα πολύ ο μιλητή και δεν υπάρχει περίπτωση να μεταφραστεί. όπω τονίζει η πρόεδρο τώρα. I'll ονομάζομαι. Είμαι σύμβουλο για την ανθρωπιστική πολιτική της Oxfam. Ξεκίνησαμε τη δράση μου το 1960. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε χιλιάδες περιπτώσεις στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ε, παροχής υπηρεσιών κτλ. Βέβαια οι προσπάθειες μας αυτές έχουν δυσκολευτεί από τις συγκρούσεις και από τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί τη βάση των ευρημάτων μετά από τις τελευταίες προσπάθειες τις οποίες κάναμε εκεί. Θα δημοσιεύσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μια έκθεση για... Σε σχέση με όλα αυτά που απασχολούν την κοινότητα και τώρα έχουμε την 50η επέτειο του του Κονγκό και η χώρα έχει 176 ε, από 182 όσον αφορά το δίκτυο τον ειδικό του ένα στα τρία παιδιά δεν μπορεί να πάει στο σχολείο υπάρχει κακή διατροφή και επίσης δεν υπάρχει και υγειονομική κάλυψη. Η κατάσταση ανθρωπιστική και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ανατολικά της χώρας είναι πάρα πολύ κακή. 5,4 εκατομμύρια έχουν χάσει τη ζωή τους από το 1998, οι περισσότεροι από αυτούς από, από θεραπεύσιμες ασθένειες και έχουμε πάρα πολλούς ε, ε πάρα, πολλούς οι οποίοι είναι άστιγοι αλλά και πάρα πολλούς πρόσφυγες από άλλες χώρες. Ξεκίνησα με αυτού του είδους ε, την εκστρατεία του FTLR στη χώρα αυτή στο Ανατολικό κογκό και ήταν οι ανθρωπιστικές συνέπειες πάρα πολύ άσχημες. 900.000 ε, ήταν αυτοί που εκτοπίστηκαν και έχουμε περίπου 1.500 οι οποίοι φωνεύτηκαν. Το 2010 έχουμε μια νέα επίθεση. Οπότε συνεχίζεται η προσπάθεια του αφοπλισμού, ε, κάποια επίσης μέτρα για διατήρηση της ειρήνης πάντως κάποιες ε, περιοχές τώρα είναι καλύτερες, ασφαλέστερες συνεχίζεται όμως ο εκτοπισμός έχουμε πάνω από 160.000 που έχουν εκτοπιστεί τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2010 έχουμε παραδιαστροπη δικαιωμάτων 246% περισσότερο στο Κύβο. Ακριβώς γιατί υπήρχαν πάρα πολλές επιθέσεις ε, οι, οι πολίτες, οι άοπλοι θα πρέπει να προστατευτεί ο πληθυσμό για να γίνει μεταρρύθμιση αστυνομία και στρατό και να υπάρχουν περισσότεροι σταθερότητα στη χώρα. Δυστυχώ, οι επαφέ με τι διάφορε κοινότητε δείχνουν ότι θεωρούν πω ο στρατό είναι αυτό που παραβιάζει με δικαιώματα. 2007-2009 έκανε η Oxfam έρευνα και 93% των όσων απάντησαν είπαν ότι το, FARDC κάνει πάρα πολλέ παραβιάσει. Και το, το ίδιο ισχύει όμως και για τον στρατό ε, όσον αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων που έπρεπε να, να ε, προστατεύουν. Ένας στους τρεις είπε ότι ο στρατός είναι η λύση, αλλά έχουν πει ότι καθημερινά γίνονται παραβιάσεις και γι' αυτό και λέμε ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση επιγόντως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει και Έχουν, έχει δοθεί νέα εντολή, νέες αποστολές του ΟΗΕ και αυτό έχει δείξει όμως ότι η εντολή αλλά και οι πόροι που διατίθενται έχουν βοηθήσει. Επίσης έχουν δοθεί πάνω από 900 εκατομμύρια ευρώ προς ε, τους φορείς που δρούν εκεί προς και την DRC 2008-2013 έχουν 561,7 εκατομμύρια ευρώ που είναι ε, μία από τις μεγαλύτερες εκταμιεύσεις σε μία και μόνη χώρα για να καλυφθούν κάποιες χώρες και να προστατευτούν ε, οι πολίτες. Διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα των ε, δύο φύλων. Και θεωρούμε ότι έτσι θα προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά συνεχώς έχουμε ομάδες παραστατιωτικών και άλλες ε, και άλλες ομάδες τα δικαιώματα, οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τι προτεραιότητε που θα τάξουμε. Η Oxfam έκανε μια έρευνα με 12 μη κυβερνητικέ οργανώσεις, 24 οργανώσεις στο Κιβού τον Απρίλιο. Είπαμε ότι πάνω από 800 έχουν φυγεί από αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. 60% των όσων απάντησαν είπαν ότι τα πράγματα φέτος είναι χειρότερα από πέρσι. Έχουμε παραβιάσει το δικαιωμάτων παντού. Ο μιλητή μιλάει όλο και πιο γρήγορα. Του το τονίζει η γιατί έτσι είναι αδύνατο να μεταφραστεί. Επομένω πρέπει να μιλήσει πιο αργά. Παντού αναφέρονται παραβιάσει των μείων δικαιωμάτων από το FDLR και άλλε οργανώσει. Απίθαργε στρατιώτε. Κατά ένα 96%. Βιασμοί, λέει λατήσεις βία σεξουαλική αυξάνεται. 20 από τι 24 ε, κοινότητες όπου κάναμε την έρευνα. Κυρίως θύματα είναι οι γυναίκες. Το 5% έλεγαν ότι είναι χειρότερα τα πράγματα από πέρσι. Νέοι επίσης, ανήλικοι. 65% είπαν ότι είναι χειρότερα. Ταπείνωση, πόνος, όλες, Ολόκληρε κοινότητε υποβάλλουν και πολλές φορές δεν βοηθούν και οι στρατιώτες που στέλνονται για να βοηθήσουν. Τα τρία τέταρτα των όσων ρωτήθηκαν είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει πολιτική λύση. Σε πολλές περιοχές. Από το 2009 έχει αποθηθεί το FTLR και έτσι όμως τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν πολύ. Η βία κατά των πολιτών ακολούθησε μετά τις στρατιωτικές επιχείρησεις στο Νότο και στο Κιβού. Όταν είχαμε την έρευνα, 99% των γυναικών και 100% ανδρών και νέων είπαν ότι τα πράγματα είναι χειρότερα από πέρσι. Λαϊλασία, ανθρωποκτονίες αυξάνονται σε σχέση με πέρσι. Είναι σαφές από τις έρευνες ότι δεν είναι δυνατόν να μετρήσουμε την ασφάλεια μόνο μέσω εχμαλώτων και μέσω των αφοπλιστέντων. Οπότε η κατάσταση επιδεινώνεται. Ζητούν λύσεις οι διάφορες κοινότητες για να υπάρχουν λιγότερες, ε, λιγότερα αντίπεινα, λιγότερες επιθέσεις. Πέρασε 1,5 χρόνος και όλες αυτές οι επιχειρήσεις δεν έφεραν τις βελτιώσεις που θέλαμε και κυρίως ανήλικοι και γυναίκες υποφέρουν από όλες τις πλευρές. Δεν πληρώνεται αρκετά, η αστυνομία δεν έχουν κοινωνική πρόνοια και ουσιαστικά και αυτοί συμβάλλουν στο πρόβλημα. Χρειάζεται περισσότερη πειθαρχία σε στρατό και αστυνομία. Και κάποια φορά η αστυνομία να προστατεύει από το στρατό. Τον κυβερνητικό. Τον DRC. Και οι διεθνεί κοινότητε να έχουν τι εξή προτεραιότητε. Πρώτον, μεταρρυθμίσει όπου θεωρούν οι κοινότητε ότι χρειάζεται. Καλύτερου μισθού στου στρατιώτε. Μόνιμε φρουρές και οργανωτική υποστήριξη ε, να αποδίδονται ευθύνε και παρά όσα έχουν γίνει, τα δύο τρίτα των όσων ρώτησε η Oxfam είπε ότι αυτό το οποίο φταίει για την καγική του στρατού είναι η χαμηλή μισθή. Ξυλοδαρμή και βιασμός. Και αυτά όλα θεωρήθηκε ότι είναι τα εγκλήματα που κάνουν οι στρατιώτες του FARDC και οι περισσότεροι από τους στρατιώτες είπαν ότι τα καταδικάζουν αλλά δεν έχουν τίποτα να φάνε. Το πρόγραμμα της USEC προβλέπει αύξηση των μισθών του στρατού. Ε, οι φταίχτες να, να εκδιώκονται από στρατό και να υπάρχει αύξηση. Έχουμε μισθούς 27 ευρω... Ε, δολαρίων. Η αποστολή του ΟΗΕ παρακολουθεί την συμπεριφορά του DRC και του στρατού τους. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλοι εταίροι. Και πάλι λέει ο Πρόεδρος στον ομιλητή ότι μιλάει πάρα πολύ γρήγορα και από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να μιλήσει πιο αργά. Και έχουμε αυτά τα σημεία ελέγχου. Και στα σημεία ελέγχου ακριβώς εκεί γίνονται οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να προστατευτούν οι πολίτε όπου δεν εξυπηρετούν τα checkpoint θα πρέπει να μετακινηθούν. Τέταρτον, πολιτικές προσπάθειες στη Ρουάντα αυτές να ενταθούν. Τέλος, ενώ συνεχίζονται επιχειρήσει, οι αρχές του Κονγκό θα πρέπει να δώσουν οδηγία σε όλους και να δοθούν εντολές να ως συνεργάτης αντίπαλης πλευράς ή άοπλη. Θα πρέπει να προστατευτεί η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια. Οι ευθύνε πέφτουν στην κυβέρνηση του Κονγκό. Αλλά θα πρέπει να βοηθήσει η διεθνή κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι το DRC να γίνει μια ισχυρή υπεύθυνη κυβέρνηση. Τώρα θα δώσω τον λόγο στην κυρία Κύρια από την Διεθνή Ομάδα Κρίσεων που είναι υπεύθυνη για το lobbying της ομάδας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας για την ακρόαση για το Κόγκο εγώ θα επικεντρωθώ στους φυσικούς πόρους και χωρίς την παρουσίασή μου σε τρία μέρη. Πρώτα απ' όλα κοιτάμε το πρόβλημα, δεύτερον κοιτάμε τη διεθνή απάντηση και στο τρίτο τμήμα κοιτάμε τις προκλήσεις για το μέλλον. Εν είδη εισαγωγής, να πω πως ε, εμείς ε, συντάσσουμε τώρα μια έκθεση για τους φυσικούς πόρους, οπότε κάνουμε έρευνα επιτόπου επ' αυτού, αλλά δεν έχουμε δημοσιεύσει τίποτα ακόμα. Το πρώτο τμήμα της παρουσίασης μου, το πρόβλημα. Είναι μια πλούσια χώρα σε φυσικούς πόρους το Κονγκό, όπως ξέρετε. Οι φυσικοί πόροι συμπεριλαμβάνουν κασιτερίτη, βολφράμιο, χρυσό, πράγματα που χρησιμοποιούνται σε τεχνολογίες όπως λάπτοπ, κινητά, αλλά ακόμα και κοσμήματα. Πολλά από τα ορυχεία είναι στρατιωτικοποιημένα από ένοπλες ομάδες αλλά και από τον στρατό. Οι εργαζόμενοι αυτοί εκεί πέρα, οι μεταλλορύχοι δουλεύουν στις σκληρές συνθήκες κάνουν με τα χέρια. Το 2001 ο ΙΕ δημιούργησε μια ομάδα ειδικών για την νόμιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και του λοιπού πλούτου του Κονγκό. Η ομάδα αυτή έκανε πολλές εκθέσεις μεταξύ 2001 και 2003 περιγράφοντας το παράνομο εμπόριο και ανέφερε εταιρείες και πρόσωπα το πάνελ αυτό αναγνώρισε την ε, σχέση μεταξύ παρανόμου εμπορίου και πολέμου. Επίσης, οι γειτονικές χώρες, Ουγκάντα και Ρουάντα, προσπαθούν να ελέγξουν τους φυσικούς πόρους και την εξαγωγή, την οποία χρησιμοποιούν για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες τους. τόνισε το πάνελ τη γενή σχέση μεταξύ οικονομικής εκμετάλλευσης, λαθρεμπορίου όπλων και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Οι εμπορικοί δρόμοι είναι μέσω Μπουρούντι και Ρουάντα 5 με 7 τόνοι χρυσού εξάγονται κάθε χρόνο γύρω στα 300 εκατομμύρια δηλαδή μέσω Ρουάντας τελικός προορισμός Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Νότια Αφρική και από Ανατολή η νόμιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων δεν προωθεί μόνο τις συγκρούσει, αλλά δεν τους επιτρέπει και να φύγουν από τις συγκρούσει. Ο αντίκτυπος είναι πολύ αρνητικός γιατί αυξάνει τη φτώχεια με το να αυξάνει τη βία και βεβαίως τις ζημιές στο περιβάλλον. Επίσης γίνεται άτυπη εξόριξη, μολύνεται το νερό και το τροπικό δάσος. Κατά το οποίο ακόμη σημαντικότερο είναι η παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων που καθιστά την διακυβέρνηση αδύνατη. Το παραεμπόριο αυτό είναι το ισοδύναμο του εμπορίου ναρκωτικών στην στο Αφγανιστάν. Φέρνει μετρητό. Οπότε αυξάνει την διαφθορά της διοίκησης και δημιουργεί μια παράλληλη οικονομία η οποία ανθεί. Και περισσότερο βεβαίως από την επίσημη. Είναι το άμεσο και μεγαλύτερο εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια σταθερότητας. Τελειώνοντας αυτό το κομμάτι της παρουσίασής μου να τονίσω πως η παράνομη εκμετάλλευση φυσικών πόρων είναι εκεί όπου συναντάται ο πόλεμος, η διεθνής οικονομία, το έγκλημα και όλες οι εμπόλεμες πλευρές εξορίσουν μέταλλα, στρατιώτες του στρατού και αντάρτες. Όλοι είναι αναμεμειγμένοι. Για το δεύτερο κομμάτι της ε, παρουσίασής μου θα εξετάσω τις διεθνείς απαντήσεις ε, οι οποίες διαφέρουν. Μία είναι η προσέγγιση δηλαδή να μποϊκοτάρουν τους εμπόρους και όχι το εμπόρευμα. Άρα έχουμε κυρώσεις κατά των εμπόρων. Δηλαδή δεν τους δίνουν βίζα και παγώνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Σε τέσσερις εκθέσεις το πάνελ του ΟΗΕ κατονόμασε αξιωματικούς στρατού, αξιωματούχους κυβέρνησης, τις οικογένειές τους που όλοι μαζί καρπώνονται τα προϊόντα της παρανομής εκμετάλλευσης. 50 εταιρείε επίσης που παραβίασαν τις οδηγίες του ΟΑΣΕ για τις πολυεθνικές. Οι εταιρείε βασίζονται στο Βέλγιο, Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία, Ισπανία κτλ. Και πουλούν όπλα στην χώρα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μια κοινή θέση το 2008 επιβάλλοντας εμπάργο όπλων, πάγωμα κονδυλίων και απαγόρευση εισόδου σε άτομα και εταιρείε που υποστηρίζουν παράνομες ομάδες ενόπλων και παραεμπόριο φυσικών πλούτοπαραγωγικών πηγών. Βεβαίω έχουμε την ε, επιβολή κυρώσεων από ασιατικές, ευρωπαϊκές και αμερικανικές χώρες. Μια δεύτερη προσέγγιση αφορά την επισημοποίηση του εμπορίου που είναι περισσότερο υπέρ της ανάπτυξης. Η προσέγγιση αυτή σημαίνει βελτίωση του διοικητικού ελέγχου για την εξόδια αλλά ε, από την άλλη πλευρά και εναρμόνιση του συστήματος στην περιοχή των μεγάλων λιμνών. Και πάλι λοιπόν οι ροές εξαρτώνται βεβαίως ε, όλα αυτά από την καλή θέληση της κυβέρνησης, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα απίθανο. Και κυρίως είπα δεν αγοράζουν τέτοια στοιχεία και μιλάμε κυρίως για μέταλλα. Οπότε απαγορεύονται αυτά τα οποία προέρχονται από περιοχές που ελέγχουν ένοπλοι και να γίνει κάτι τέτοιο υποχρεωτικό για τις εταιρείε ηλεκτρονικών πίεση σε εταιρείε από το κοινό για να μην χρησιμοποιούν τέτοια μέταλλα και να κατονομάζουν τις εταιρείε. Και το σχετικό νομοθέτημα είναι ακόμα στο Κογκρέσο. Και υπάρχει βεβαίως το στρατηγικό σχέδιο δράσης το οποίο έχει εγκριθεί. Με συγχωρείτε αγαπητή μου κυρία λέει πρόεδρος ε, έχουν περάσει 8 λεπτά και είστε ακόμα στη μέση του δεύτερου μέρους. Ε, πρέπει να συζητήσουμε κιόλα κάποτε. Και στην περίπτωση των ΗΠΑ το στρατηγικό σχέδιο δράσης για τα μέταλλα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών το Μάρτιο. Τα προβλήματα είναι πάλι η δυσκολία χαρτογράφησης αυτοσχεδίων μεταλλίων και η μη συμπερίληψη αυτών υπό τον έλεγχο του στρατού και βεβαίως το ότι δεν υπάρχει δέουσα επιμέλεια. Οι προκλήσεις λοιπόν για το μέλλον. Η διεθνής κοινότητα συζητάει το τι πρέπει να γίνει. Η άποψή μας είναι πως δεν έχει συζητηθεί το τι μπορεί να γίνει στην περιοχή των μεγάλων λιμνών. Κατά την άποψή μας, υπάρχουν δύο πολύ προβληματικές πτυχές. Η έλλειψη συντονισμού, οι βιομηχανίες, οι, οι επιστήμονες διεθνείς οι οργανισμοί, το κοιτάω καθένα από τη δικιά του σκοπιά. Δεν υπάρχει συντονισμός. Και δεν ξέρουμε αν είναι και συμβατές αυτές οι προσεγγίσεις. Αυτή τη στιγμή είπα, είναι οι πιο προχωρημένες και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ. Δηλαδή να γίνει υποχρεωτική ιδέουσα επιμέλεια. Το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι η έλλειψη πολιτικού ρεαλισμού. Δηλαδή απαιτείται περιφερειακή λύση γιατί περιφερειακό είναι το εμπόριο μετάλλων. Γιατί πρόκειται για διεθνές εμπόριο όμως και η προσέγγιση αυτή η περιφερειακή είναι λανθασμένη. Με συγχωρείτε λέει πρόεδρος, ε, αργείτε σε δύο λεπτά και τελείωσα. Λοιπόν και επειδή το άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης ε, από τις κυβερνήσεις της περιοχής των μεγάλων λιμνών. Μάλιστα σας ευχαριστώ. Νομίζω πως μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Ο κύριος Τάνοκ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι η κατάσταση και η Δημοκρατία του Κονγκό είναι ανησυχητική. Εγώ συμμετείχα σε μια συζήτηση στο Στρασβούργο. Στην τελευταία ολομέλεια. για την δολοφονία του υπεραστή αυτού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μπισκάλντι, νομίζω το ανέφερε, είναι κάτι το οποίο εγώ λέω εδώ και καιρό. Με βάση την ε, επιτυχία της διαδικασίας Κιμπάλη για διαμάντια από πολέμους, πώς χρειάζεται να δούμε κάτι το ευρύτερο. Πέρα από τα διαμάντια, να δούμε κάτι και για μέταλλα, ειδικά χαλκό και διάφορα άλλα σπάνια. Ειδικά από κάποιες ε, περιοχές Αφρικής όπου γίνονται επιχειρήσεις και από τον τακτικό στρατό και τις παραστρατιωτικές ομάδες και πολλές κατηγορίες ανταλλάσσονται όπου μιλάμε η διαφθορά έχει φτάσει στα όρια της κλεπτοκρατίας ε, επί Μομπούτου. Ε, Πώς λοιπόν έτσι μπορέσουμε να είτε να έχουμε επέκταση της διαδικασίας Κιμπάλη ή μια νέα επιτροπή υπό την ηγεσία της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βεβαιώσει την προέλευση των μετάλλων. για να μην πηγαίνουν τα λεφτά είτε στη διαφθόρα είτε σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ μου υπενθύμησαν πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε πράγματι ένα ψήφισμα για την παρανομή εκμετάλλευση των πόρων στο Κονγκό και ζήτησε από τα κράτη-μέλη να ερευνήσουν τις εταιρείες της Ένωσης που αναφέρονται σε εκθέσεις του ΟΗΕ του 2002 και 2003. Ο κύριος Γκέρεντς Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με εντυπωσίασαν πάρα πολύ τρεις ε, εισηγήσει που ακούσαμε. Και η όσα είπε ο πρώτος από τους ομιλητές όσον αφορά αυτά τα εγκλήματα και τα οποία κάθε που γίνονται ε, συγκροτούμε με κάποια διεθνή επιτροπή και οπότε δεν πρωτοτυπούμε. Κάθε φορά που υπάρχει ένα συμβάν γίνονται τα ίδια. Αντιδρούμε τον ίδιο τρόπο. Τον ίδιο τρόπο, τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο. Έχω όμως βάσει το άρθρο 8 της συνθήκης Κοτονού. Εκεί θεσπίζεται ένας προληπτικός μηχανισμός αποδεκτός από όλα τα μέρη της ΑΚΕ που ακριβώς συμφώνησαν να υπάρχει μια αμερόληπτη διεθνής επιτροπή. Αυτή είναι η αρχή. Δεν γίνεται να κάνουμε αυτό που προβλέπει το άρθρο 8. Δεύτερον, η συνθήκη Κοτονού ήταν εφορμή να πιεστούν οι χώρε τη Αφρική με Ευρωπαϊκή για να δεχθούν το να ληφθεί υπόψη περισσότερο ιδιωτικό τομέα και η κοινωνία των πολιτών. Αναφέρθηκαν ένα σωρό στοιχεία σχετικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια συνειδητοποιημένη διεθνή κοινότητα που να μπορεί να λειτουργήσει. Δεν ήταν εύκολο να πέρασει αυτή η ιδέα ε, χρειάστηκε να πιέσουμε το 2000 ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και στάθηκαν πάρα πολύ δύο χώρες της Αφρικής αλλά τελικά δέχτηκαν αυτό που προτείναμε τώρα όσον αφορά την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και επ' αυτού θα έπρεπε να εκθέσουμε τις προτάσεις μας ως Επιτροπή, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και από ό,τι διαπιστώνουμε ο ιδιωτικός τομέας ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί όσο θα έπρεπε. Ξέρω ότι η Επιτροπή έχει ενεργοποιηθεί για να δημιουργηθεί μια συνένεση, αλλά τα πράγματα ακόμα είναι αρκετά πρωτόγωνα. Αυτό θα σας πω για να προβληματιστούμε σε σχέση με αυτά που ακούσαμε, για να τα λάβουν υπόψη οι εισηγητές μας, αλλά και εμείς. Ευχαριστούμε, κύριε Γκέρνς. Πάρα πολύ σωστή αυτή η πρόταση που πηγάζει από το άρθρο 8 της Συμφωνίας Κοτονού. Βέβαια, η ισομερή και η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως είναι ε, το κατάλληλος τόπος τόσο ώστε να συζητήσει κανείς για μια τέτοια αμερόληπτη επιτροπή. Είναι αλήθεια όμως ότι τα ίδια κάνουμε σε κάθε περίπτωση και κάποια φορά χρειάζεται να υπάρχουν διαφοροποιήσει και να αναρωτιέται κανεί ποια είναι κάθε φορά πιο δόκιμη λύση. Η επόμενη μιλήτρια είναι η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπω είναι μεγάλη υπογοήτευση ματέως αυτή η υπόθεση ε, του DRC το 2006 προσπαθήσαμε με μια αποστολή να βοηθήσουμε για να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσον η αποστολή έφερε αποτελέσματα. Τα δικά μου συμπεράσματα είναι ότι όλα όσα κάναμε δεν βρήκαν απόκριση από στη DRC. Άλλοι έχουν κάποια κίνητρα, έστω και δύο τελεία, άλλοι δεν ενδιαφέρονται. Το EDF μας δίνει τόσα πολλά χρήματα, τόσα που αποδέκτης τους στην ίδια. Όμως, αυτοί που ασχολούνται με την κοινωνία ο κ. Μουκέλα, μα λένε ότι δεν παίρνουν εκείνοι τίποτα από αυτά τα χρήματα. Δεν στηρίζονται οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Όπω μα είπε ο κ. Μουκέλα. Μ' ακούσαμε τον κύριο Γκότσελκ μας είπε ότι ότι από κάποιες αποστολές κάτι προέκυψε. Όμως Τελικά δηλαδή δεν καλύπτονται αυτά τα οποία πραγματικά θα έπρεπε να καλύπτονται. Και επομένως είναι πάρα πολύ μικρή αποτελεσματικότητα αυτών των κονδυλίων. Άρα βεβαίως και χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Ε, αλλά δεν είναι μόνο οι μεταρρυθμίσεις του στατού και της αστυνομίας. Χρειάζεται να αναβαθμιστούν όλες τις παραγωγές δυνατότητες της χώρας. όλη η χώρα για να μπορούσουμε να δούμε κάποια διαφορά. Οι προσπάθειές μας δεν πιάνουν τόπο καθόλου. Δηλαδή και τελικά ούτε προστατεύουν αυτούς που θα έπρεπε. Γι' αυτό βλέπουμε ότι δολοφονούνται αυτοί οι αγωνιστές. Περίπτωση Αγκάντα. Νομίζω ότι το, το DRC το ίδιο παρέπεμψε την περίπτωση, την υπόθεση αυτή στο Διεθνές Δικαστήριο. Δεν τον παρέδωσε όμως. Και μάλιστα του έδωσε και προαγωγή. Και κανείς δεν κάνει τίποτα, κανείς δεν το λέει αυτό. Πήγα στην κουμπάλα women and, and as it had been highlighted and everybody in the Great Lakes area it's, it's a disaster. Είδαμε τη τραγωδία επικρατήσει στην Μίζωνα περιοχή των ε, μεγάλων λιμνών ε, είχαμε ένα σωρό ακροάσεις είχαμε το ψήφισμα για τον αγωνιστή που σκοτώθηκε αλλά είναι πάρα πολύ αναποτελεσματική η δράση μας δηλαδή για το 8, για το άρθρο 96 της ΑΚΕ πάρα πολύ λίγα γίνανε κυρίως, κυρίως για το Κονγκό Τίποτα δεν γίνεται. Και το πιο σημαντικό, εκτός από τις μεταρρυθμίσεις, είναι το τι θα γίνει με τους φυσικούς πόρους. Μα όλοι στη συνέλευση ΑΚΕ, τότε το 2008 που συναντηθήκαμε στην Παππούνια Νέα Γουινέα, όλοι ήμασταν και το είπαμε ότι θα πρέπει να κατονομαστούν, να κατηγορηθούν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές, πολυεθνικές, όλες όσες εκμεταλλεύονται την κατάσταση εκεί, όσοι συμμετέχουν σε αυτόν τον φαύλο κύκλο. να κερδίσουμε την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Ούτε έγινε τίποτα και από την πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα αυτό νομίζω πρέπει να κάνουμε. Έχει δίκιο ο κυρία Μπισκάλτη. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνει η Αμερικάνια. Όχι, όχι, το ένα ψήφισμα μετά τον άλλο. Το ένα ψήνει το άλλο και κανείς δεν δίνει δεκάρα. Αποστολή στο Κονγκό και οι άξονες δράσεις θα είναι πρώτα-πρώτα σεξουαλική βία περιοχή των μεγάλων λιμνών, λιμνών και δεύτερον εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Ε, να σκεφτούμε συγκεκριμένους τρόπους για να ξεσκεπάσουμε τους υπεύθυνους αυτής της τραγωδίας. Δεν χρειάζεται να ξαναφεύγουμε τον τροχό. Κυρία Μπισκάλντι, πέστε μας δύο λόγια όσον αφορά τον ρόλο της Κίνας στο Κονγκό. Γιατί ένα από τα πιο απαράδεκτα το οποία έχουν γίνει, φυσικά και η Κίνα εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους και βέβαια σε, από πλευρά ανάπτυξη ε, όλο και κάτι ωφελούν αυτά για το Κονγκό. Όμω οι συμβάσει αυτέ είναι λεόντιε, τερατώδει. Θα πρέπει να συμφωνείτε τι γίνεται, πού γίνεται σχολεία, δρόμοι. Και υπάρχει σιωπή, ομερτά από πλευρά δική μα, από πλευρά τη Παγκοσμία Τράπεζα, για ένα σωρό συμβάσει που είναι αρνητικέ, επιζήμιε. Ε, είναι καθαρά ε, απεικιοκρατική αυτή η εκμετάλλευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε έτσι πολύ ωραία, αναλυτικότατα. Τα θυμόμαστε την πρότασή σας. Ναι. και αυτό το οποίο είπατε για τη βία κατά των γυναικών και την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι κάτι που είναι πάντα στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας και είναι ενισχυτικό αυτό το οποίο συμβαίνει οι οικογένειες του κυρίου Τσεμπάγια και των συναδέλφων του απειλούνται αν κατάλαβα καλά επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τόμσκης, και μετά θα ζητήσω από την Κομισιόν να παρέμβει. Κύριε Τόμσκης, ναι αγαπητοί συνάδελφοι, μία παρατήρηση έχοντας ακούσει τα πολύ ενισχυτικά αυτά νέα και σχόλια θα ήθελα να πω κάτι. Εγώ παρακολουθώ την ακαδημαϊκή συζήτηση για τον συστηματικό βιασμό των γυναικών στο Κονγκό και αυτό το οποίο είναι πραγματικά ανησυχητικό είναι πως κάποιοι άνθρωποι στα πανεπιστήμια το ορίζουν ως κάτι το πολιτισμικό. Δηλαδή αυτός ένας, ένας ε, πολιτισμικός ε, ε, ρελατιβισμός που είναι σοκάρι. Εντάξει, να σκεφτούμε τι γίνεται στο Κονγκό. Αντιλαμβάνω πώ θα υποφέρει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ των διαφορετικών πτυχών των φαινομένων. Και όμω, γεγονό παραμένει πω πουθενά στον κόσμο οι ζωέ των γυναικών δεν απειλούνται περισσότερο από τι χώρε αυτέ. Από τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Γι' αυτό αυτές οι μορφές μισογενίας, μισογενισμού, με απαιτούν να δραστηριοποιηθούμε. Πρέπει να ορίσουμε μια σωστή γλώσσα κιόλα, γιατί καμιά φορά οι όροι που χρησιμοποιούμε μοιάζουν ξεφτισμένοι και δυσλειτουργικοί για να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, μιλάμε για σεξουαλική βία και η λέξη δεν περιγράφει το φαινόμενο. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω να έχουμε μια σωστή ορολογία όταν ε, μιλάμε για την άρνηση της αξιοπρέπειας των γυναικών. Έχω για το επίπεδο αυτό της, μιλάμε, πλησιάζει το επίπεδο της γενοκτονίας, συστηματικής καταστροφής, αξιοπρέπειας και ζωής των γυναικών. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε κάτι. Ίσως για πρώτη φορά στην ε, σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας οι γυναίκες εξοντώνονται ηθικά και σωματικά. Ευχαριστώ κύριε Τιόντσκης. Η Ελιζαμπέτησο από την Γενική Διεύθυνση την Αρμόδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. <clears throat> Θα ήθελα σύντομα να αντιδράσω σε ορισμένες από τις παρεμβάσεις οι οποίες προηγήθηκαν. Είναι προφανές ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναπόσπαστο τμήμα των αξιών της Ένωσης και είναι θέμα το οποίο προωθεί πάντα στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο. Στο Κογκό η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ κακή. Πώς να αγνοεί κανείς ε, τις ε, καταστάσεις που ακούσαμε προηγουμένως που πράγματι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, σεξουαλική βία, βία εναντίον των παιδιών, βία εις βάρος των δημοσιογράφων <clears throat> και των αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπροστά σε όλα αυτά θα πρέπει να καταγγείλουμε την κατάσταση και να βάλουμε στην ημερήσια διάταξη τα θέματα των γυναικών και των παιδιών στην Δημοκρατία του Κόγκο. Είναι απαραίτητο να, δώσουμε τις, να πάρουμε τη σκητάλη από την κοινωνία των πολιτών, η οποία προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση εκεί όπου η εξουσία δεν είναι σε θέση να <clears throat> αλλάξει τα πράγματα. Και εδώ κανένας δεν αναφέρθηκε στο κοινοβούλιο, το οποίο και αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί. Πιστεύουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά και θα πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλους οι οποίοι πιστεύουν σε αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κατάσταση και προσπαθούν να δράσουν συντονισμένα. Σχετικά με τις συστάσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, θα ήθελα να πω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάντα σε μια υψηλή θέση στα πλαίσια του διαφθομένου πολιτικού διαλόγου θέλουμε, που θέλουμε να προχωρήσουμε και να εμβαθύνουμε μέσω του άρθρου Ακόμα και αν τα θέματα αυτά συζητώνται συχνά με τις αρχές της χώρας, είναι σαφές ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η θέση τους. Για την κοινωνία των πολιτών θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μέσω των ταμείων του ΦΕΔ και μέσω άμεσων βοηθειών. Τα πέντε τελευταία χρόνια έχουμε συνεργαστεί με 50 οργανώσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας που βοηθούν τα θύματα, που πλαισιώνουν τα παιδιά που είναι εγκαταλελειμμένα και που ενισχύουν τις τοπικές αρχές. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε σημαντική πρόοδο είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς το πλαίσιο των προβλημάτων και να βρει τις διαφορετικές δράσεις που θα βοηθήσουν να καλυφθούν οι προτεραιότητες. Ξέρουμε ότι για πάρα πολύ καιρό είχε διαλυθεί πλήρως το κράτος δικαίου η βία που είχε χαρακτηρίσει την εποχή αυτή συνεχίζει δυστυχώς να παραμένει σε ορισμένες περιφέρειες. Οι προσπάθειες ανοικοδόμησης του κράτους στο Κονγκό και η πολιτική μετάβαση αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα και απαιτούν προσπάθειες οι οποίες δεν μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμες. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προϋποθέτει την πολιτική βούληση αλλά και την κυριαρχία του δικαίου και εδώ υπάρχουν πολλά να γίνουν. Υπάρχει τρομερό έλλειμμα σε σχέση με την παρουσία του κράτους και την αντικειμενικότητα της διοίκησης που είναι ανεπαρκέστατη και πηγή ανασφάλειας. Και η μάστιγα της ατιμορρησίας η οποία πάντα σοβεί. Η δικαιοσύνη είναι ελληματική όχι μόνο στην παραγωγή της ίδιας της δικαιοσύνης αλλά και στην δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Τέλος και η ποινική διαδικασία από την αστυνομία μέχρι τη δικαστική εξουσία είναι απαράδεκτη για να μην μιλήσω για τις φυλακές. Η διάρκεια των συγκρούσεων έχει οδηγήσει σε περίπλοκες καταστάσεις σε επίπεδο ε, δυνάμεων τήρησης της τάξης, των οποίων η συγχώνευση είναι απαραίτητη σήμερα περισσότερο από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαρωτώνται τι πρέπει να γίνει σε σχέση με την εικόνα αυτή η δημοκρατία του Κονγκό έχει βρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα επικοδομητικό εταίρο, διότι πρέπει να είναι κανείς επικοδομητικός και όχι μόνο καταγγελτικός. Οι επαφές θα πρέπει να συνεχιστούν με στοχευμένο τρόπο. Θα πρέπει επίσης να στηρίξουμε το τέλος των συγκρούσεων, γιατί ε, προφανώς το δίκαιο δεν μπορεί να υπερισχύσει όταν υπάρχουν ανοιχτές συγκρούσεις όταν υπάρχουν μάχες αυτές στοιχειοθετούν ανοιχτές απειλές για τους πληθυσμούς. Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν στην ανοικοδόμηση σύμφωνα με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης της Κινσάσα. Πέραν από την ηλική ανοικοδόμηση απαιτείται και η ανοικοδόμηση του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και της αστυνομίας από το 2004 οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ιδιαίτερα σημαντικές στον τομέα της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. 100 εκατομμύρια ευρώ έχουμε διαθέσει προς την κατεύθυνση αυτή σε σχέση με τον εξυγχρονισμό του δικαϊκού συστήματος, την βοήθεια στα θύματα και την βελτίωση των θεσμικών δομών και οργανώσεων και την κατάρτιση των αστυνομικών και δικαστών. Φυσικά υπάρχουν και βοήθειες διμερείς από τα κράτη-μέλη και ε, υπάρχουν και δύο διεθνείς δράσεις παρούσες στο Κονγκό για να βοηθήσουν να διοχετευθεί σωστά η ευρωπαϊκή βοήθεια. Αυτά όμως δεν θα πρέπει να εκλειθούν σαν μια καταγγελία πολιτική. Κοιτάξτε, συγγνώμη, μια στιγμή διακόπτει η Πρόεδρος για μια ακόμη φορά μου ζητούν ότι εφόσον διαβάζετε τόσο γρήγορα δεν μπορούν να σας διευμηνεύσουν, δεν σας παρακολουθούν γενικά οι διευμηνείς. Είναι καλύτερα φυσικά να μην διαβάζει κανείς τα κείμενά του, αλλά εφόσον τα διαβάζει ας τα ομιλεί αργά. Λοιπόν, οι προσπάθειες αυτές συνδυάζονται με τις προσπάθειες της διμερής των κρατών μελών και των δύο διεθνών αποστολών που είναι παρούσες στο Κονγκό και βοηθούν με σημαντικό τρόπο στην διοχέτευση της ευρωπαϊκής βοήθειας. Είχα μιλήσει για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την αποκατάσταση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Δεν θα πρέπει όλα αυτά να εκλειφθούν σαν πολιτικές καταγγελίες. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες μπροστά στην πολιτική τάξη του Κονγκό και δυσκολίες και για τη στάση την οποία θα πρέπει να κρατήσει η διεθνής κοινότητα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Τίσο. Μου υπενθύμησαν ότι όταν πήγε η Υπουργό Κλίντον στο Κονγκό τον Αύγουστο του 2009 πήγε με ένα πρόγραμμα 70 εκατομμυρίων ευρώ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας. θα εκπαιδεύσει γιατρούς, θα βοηθήσει τα θύματα. Γενικά έχουν πάρει μέτρα δηλαδή, προσπαθούν να βοηθήσουν με συγκεκριμένα επιτόπου μέτρα και αναρωτιέμαι αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δει τα θέματα αυτά στη βάση τους, στο επίπεδο στο οποίο προκαλούνται. Και προφανώς το θέμα είναι ότι και η συνάντηση, η διακοινοβουλευτική ΕΟΚΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ θα πρέπει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει να μιλήσουμε και με τον κύριο Μισελ, ο οποίος δεν θα πρέπει να αγνοήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στις συζητήσεις που έχει για το Κογκό. Αυτά. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους τρεις ομιλητές που πήραν το λόγο να κάνουν ε, κάποια σχόλια ή κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα οποία ακούστηκαν προηγουμένως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους κυρίους βουλευτές που πήραν το λόγο. Συμφωνούμε ως προς την καταδίκη αυτών των ενεργειών και την αποστολή μιας Επιτροπής Έρευνας. Επιτόπου τώρα, οι κατευθυντήριες γραμμές, οι σχετικές με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με την προστασία αυτών που τα προασπίζονται, δεν εφαρμόζονται σωστά. Δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά. Δεν υπάρχει παρακολούθηση των δικαστικών διαδικασιών δεν υπάρχει πολιτική στήριξη προς αυτούς οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι προσπιζόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεν υπάρχει και οικονομική στήριξη στις πλέον ανεξάρτητες οργανώσεις οι οποίες έτσι καθίστανται φυσικά και οι λεγότερο θεσμικές, οι πιο εκτεθειμένες και οι πιο εύθαστες απέναντι στην κρατική καταστολή. Σχετικά με τον πολιτικό διάλογο τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέγει ότι ο πολιτικός διάλογος υπάρχει. Εμείς δεν τον βλέπουμε, δεν τον αισθανόμεθα. Ποιος μπορεί να μας πει σήμερα το πότε και πού έγινε η τελευταία συνάντηση του πολιτικού διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 8 ποια ήταν η μερίσια διάταξη του διαλόγου αυτού. Τι απάντησαν στις αιτιάσεις μας ε, οι αρχές. Εμείς προσπαθούμε να λειτουργήσουμε σαν αντιεξουσία για να βελτιώσουμε έστω και κατ' λίγο την κατάσταση αυτή. Κανένας δεν μας πληροφορεί, κανένας δεν μας ενημερώνει, κανένας δεν μας διαβουλεύεται. Προφανώς αναφορές στην κοινωνία των πολιτών γίνονται η οποία όμως δεν είναι παρούσα εκεί όπου δίδονται οι μάχες για την βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν τμήματα σε εισαγωγικά της κοινωνίας των πολιτών η οποία υπακούει πιστά στην εξουσία. Έχω ζήσει το σύστημα αυτό και συνεχίζω να το βιώνω επί τόπου. Εξακολουθώ να πιστεύω οι ανεξάρτητες οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών δεν ε, ακούγεται η φωνή τους. Να κάνετε μία αποστολή, όχι μόνο όμως στο θέμα της βίας της βάρος των γυναικών, και αυτό μας απασχολεί φυσικά. Και όχι μόνο σε σχέση με την κατασπατάληση των φυσικών πόρων της χώρας αλλά σε σχέση με το πώς διατίθενται όλα αυτά τα εκατομμύρια εκατομμυρίων τα οποία διατίθενται στη χώρα αυτή. Για τον κύριο Ντόνσκης. Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες είναι τα πρώτα βήματα, θύματα, συγγνώμη, της βίας και της ατιμορρησίας. Το λέμε αυτό, το καταγγέλουμε αυτό σχετικά με τον πολιτιστικό τρόπο σχετικοποίησης. Ε, η οργάνωσή μου και τα μέλη της έχουν προσπαθήσει να λειτουργήσουν σαν αλυσίδα ενημέρωσης κατά αυτής της κατάστασης. Αυτά είχα να πω πρόεδρε προς το παρόν κάποιες παρατηρήσεις και απαντήσεις σε αυτά τα οποία είπαν οι προηγούμενοι μέλη του Κοινοβουλίου. Πάρα πολύ πολύτιμα όλα αυτά για να τα ξέρουμε. As a follow-up of this hearing, uh, I'm going to contact the ambassador and I'm going to... Και τι θα μιλήσω και με τον πρέσβη και θα μιλήσω συνήθως μας είπατε ίσως να στείλω και στην αντιπροσωπεία της Ένωσης στη χώρα μια επιστολή γιατί θα πρέπει τα πράγματα πάνε καλύτερα από ό,τι μας είπατε. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Για να μας πει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν ε, θεωρεί ότι αυτά όλα τα θεμητά αιτήματα του κύριου Κακούλα ε, είναι δυνατόν να μας οδηγήσουν σε μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών στο Κονγκό. Και έτσι οι αντιπροσωπείες στην Κινσάσα να οργανώσουν επιγόντως μία συνάντηση με τις αρχές για να βρεθούν κάποιοι μηχανισμοί προειδοποίησης για την προστασία των όσων μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι λέτε, Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. σιγά σιγά υλοποιούμε τις καθημερινές γραμμές για την προστασία των όσων αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια τοπική στρατηγική ξεκίνησε τον Μάρτιο. Σύμφωνα με αυτήν υπάρχουν διαφορετικοί μηχανισμοί. Εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ δηλαδή αυτών και των ε, πρέσβεων για την περίπτωση επίγοντος και υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης σε περίπτωση που υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα, κάποιες περιοδικές επισκέψεις στις μη κυβερνικούς οργανισμούς και συναντήσεις με αυτούς τους αγωνιστές για τα δικαιώματα. Γι' αυτό επιδέχεται βελτίωση. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε τώρα πρόσφατα το Μάρτιο και όλα αυτά γίνονται εις συντονισμό με τους εκπροσώπους του ΟΗΕ. Εδώ και πολύ καιρό συνεργαζόμαστε με τον ΟΗΕΓΙ. Όσον αφορά το άρθρο 8, εδώ έχουμε αυτές τις καθεντήρες σε σχέση με το πώς θα επικαλεστούμε, πώς θα δράσουμε δυνάμει του άρθρου 8 με τον πιο ευέλικτο τρόπο σε σχέση και με την Διεθνή Οργάνωση για Ανθρώπινα Δικαιώματα ότι θα πρέπει δηλαδή να Διαβουλαυτούμε με τους σχετικούς φορείς των ανθρώπινων δικαιώματα πριν προχωρήσουμε σε αυτή την πολιτική συμφωνία που θα πρέπει το άρθρο 8 βέβαια να ενεργοποιηθεί αλλά όμως θα πρέπει να γίνει και πολιτικός διάλογος με τις αρχές για να μπορέσουμε να έχουμε ε, μια ε, μερίσια, δηλαδή, χάρτη πορείας που να είναι αποδεκτός από τις αρχές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούμε ότι αυτή η στρατηγική έχει αποφασιστεί τον Μάρτιο, αλλά τι γίνεται. Μπορούμε να, να, να δούμε ότι όντω υπάρχει ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει επίση. Όπως γνωρίζετε πρόεδρε, προσπαθήσαμε με την Ισπανική Προεδρία να οθήσουμε την υλοποίηση των κατευθυρίων γραμμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έγιναν επαφές με τις αντιπροσωπείες εκεί, με τις πρεσβείες όλες αυτές οι στρατηγικές όλα αυτά που έγιναν και όσον αφορά την εκστρατεία ευαισθητοποίησης Είπαμε να γίνει αυτό όπου υπάρχουν στρατηγικέ. αλλά ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει. Δεν έχει γίνει δημοσίευση ακόμα γιατί καταλαβαίνετε είναι χώρε με δύσκολες συνθήκες όσον αφορά αυτή την ενημέρωση. Υπάρχει πρόβλημα ακόμα και με το περιεχόμενο της εκστρατείας σε σχέση με τις αρχές. Ε, είναι δύσκολη υπόθεση η προστασία των αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, ε, αφενός έχουμε τη στρατηγική και αφετέρου έχουμε αυτή την στρατηγική της συνειδητοποίησης ότι υπάρχει πολιτική τέτοια. Ξέρουμε ότι πρέπει να προστατευτούν αυτοί οι αγωνιστές. Όχι, δεν λέμε να δημοσιεύσετε τις πληροφορίες για το τι γίνεται Θα πρέπει κάποια στοιχεία όμω να δημοσιοποιηθούν. Έχουμε εμείς και τον κανονισμό για την προσβασιμότητα στα επίσημα έγγραφα. Οπότε... Μπορεί κάποιος να δει πώς έχουν προχωρήσει αυτές οι εκστρατείες ενημέρωσης. Ευχαριστώ που μου δίνετε πάλι το λόγο. Θα είναι σύντομη έτσι, και θα κάνω κάτι σχολιάκια για την διαδικασία Κιμπάλη και τον ρόλο της Κίνας. Και θα συναντήσω προσωπικά τον κύριο Προβουλευτή αφού συμβουλευτώ τον αναλυτή μας επιτόπου για να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες θα έλεγα πως ε, σε γενικές γραμμές οποιαδήποτε λύση σε σχέση με την ε, παράνομη εκμετάλλευση φυσικών πόρων θα πρέπει να ελεγχθεί Δηλαδή, οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να βασίζεται σε μια αξιολόγηση των αναγκών σε πολιτικό πλαίσιο και να δούμε τι είναι εφικτό στο πλαίσιο του Κονγκό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους φυσικούς πόρους, αλλά είναι και ένα μάθημα που μάθαμε από το τομέα, τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας. Και αυτό γιατί κατά κάποιον τρόπο η παραοικονομία είναι δείγμα του ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει τους νόμους εθνικούς και διεθνείς και αυτό δεν θέλει να το κάνει το εμπόριο και η οικονομία αυτή η παράνομη ανθεί περισσότερο από την επίσημη οικονομία. Και υποφελούνται έτσι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ειδικά τώρα σε σχέση με κάποια σχόλια που κάναμε για τον πολιτικό διάλογο και το άρθρο 8, ενδιαφέρον θα είναι να δούμε τη συζήτηση περί παρανόμου εμπορίου πρώτων και το τι μπορεί να γίνει με το άρθρο 8 κατά τρόπον ώστε οποιαδήποτε λύση πολιτική ή έργο της Ένωσης να ελέγχεται όσον αφορά και την πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπισκάλντι για τις εξαιρετικές σας προτάσεις. Κύριε Κότσολκ, θέλετε τον λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε έτσι γρήγορα, συνειδητοποιώ ε, πως παρουσίασα πολλά στατιστικά στοιχεία και είναι δύσκολο να ακουστούν ε, όταν μιλάω τόσο γρήγορα. Απλά θα ήθελα να πω πως μία έκθεσή μας υπάρχει στα έγγραφά σας και άλλη μια έκθεση πιο πρόσφατη με τίτλο «Πρώτα τα γυναικόπαιδα στα μέτωπα». Ε, θα δημοσιευθεί την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε θα μπορέσετε να δείτε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία και συστάσεις εκεί. Και κάτι άλλο γρήγορα. Να συμφωνήσω με τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν ε, για το ότι πραγματικά οι πόροι που αφιερώνονται δεν επαρκούν. Δηλαδή το να δούμε τι ότι έχει επιτευχθεί παρά τους πόρους αυτούς ε, πραγματικά τιμά όσους είναι εκεί πέρα αλλά καθώς σε συζητάμε τώρα πρέπει να ξαναδούμε τις ε, δεσμεύσεις των κρατών μελών. για να μπορούμε να κάνουμε αυτή την πολύ σημαντική συνεισφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκότ Σάλκ. Τελευταία ομιλήτρια η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Πράγματι ήταν συνάντηση σημαντική αυτή η συνάντηση. Η κατάσταση είναι τραυματική για όλους στο Κονγκό. Φυσικά και οι δολοφονίες των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης, οι ταπεινώσεις που υφίσταται ο πληθυσμός βλέπουμε ότι η κατάσταση σε επίπεδο σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαράδεκτη. Υπάρχει έντονη καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα για την κατάσταση των γυναικών στη χώρα αυτή. Ο πληθυσμός της υποφέρει, εξολοθρεύεται εν πολλής Είχε πάει η κυρία Κλίντον, είχε κάνει μια περιοδία σε κάποιες περιοχές απομεμακρυσμένες, φάνηκε ότι υπήρχαν κάποιες βελτιώσεις, τώρα η κατάσταση έχει επανέλθει δυστυχώς στην άσχημη κατάσταση που ήταν πριν. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε αρκετά διεθνή μέσα. Η κυρία Γκόμες αναφέρθηκε σε αυτά τα μέσα Έχουμε συζητήσει ήδη με τον Επίτροπο Ντεχούχτ για την κατάσταση των γυναικών. Ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε και από την Ανωτάτη Εκπρόσωπο για τα εξωτερικά θέματα και από την Επίτροπο για την, τον Επίτροπο για την Ανάπτυξη να συζητήσουν μαζί μας μια ουσιαστική στρατηγική για μια κατάσταση η οποία δυστυχώς χειροτερεύει. Φυσικά και πρέπει να συνεννοηθούμε και με τα Ηνωμένα Έθνη. Είχαμε προβλήματα και με την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών. Ξέρετε ότι συστηματικά προέβαιναν σε βιασμούς γυναικών οι στρατιώτες της δύναμης αυτής της ειρηνευτικής. Πήρε τα κατάλληλα μέτρα από ό,τι φαίνεται η διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών εις βάρος αυτών των στρατιωτών οι οποίοι είχαν σταλεί εκεί για να προστατεύσουν τον πληθυσμό και όχι για να συμμετέχουν στην <clears throat> καταστροφή του. Θα πρέπει να ζητήσουμε επίσης και από τους εκπροσώπους του Διεθνούς Δικαστηρίου να τα συζητήσουν τα θέματα μαζί μας για να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της ε, ατιμορρησίας που δεν πάβει να αλλάζει δυστυχώς. Σύνεπως θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο δραστήριοι στον συγκεκριμένο τομέα από ό,τι μέχρι τώρα. Να είμαστε προσεκτικοί για τις επιθέσεις εις βάρος ε, της κοινωνίας των πολιτών και στο τέλος, τέλος να μιλήσουμε και για πιθανές κυρώσεις αν αυτό είναι απαραίτητο. Ελπίζω λοιπόν μετά από τις ε, διακοπές να επανέλθουμε στο θέμα πιο συστηματικά. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τους προσκεκλημένους. Εύχομαι θάρρος και κουράγιο και δύναμη σε όλους, ιδιαίτερα εσάς που έρχεστε από την χώρα αυτή. Αυτά τα οποία είπατε και τα αιτήματά σας κρίνονται απολύτως λογικά και μετριοπαθή και ελπίζω να γίνουν δεκτά. Uh, um, Θεωρώ λοιπόν πως θα πρέπει να μιλήσουμε και με τον κύριο Μισελ, τον συμπρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ για να ακολουθήσει κάποιες από αυτές τις προτάσεις που ακούστηκαν εδώ μέσα. Έτσι ώστε η επόμενη κοινοβουλευτική της σας αν είναι Σε Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Και την κατάλληλη στιγμή ε, μπαίνει ο κύριος Μπροκ, ούτε νωρίς έχει έρθει ποτέ του, ούτε όμως και αργά. Έλμαρ, παίρνα. Κάτσε κάτω που θες, Έλμαρ. Λοιπόν, καλώς ορίζω εδώ τον συνάδελφο, τον κύριο Μπροκ, για να μας εξηγήσει τον τελικό συμβιβασμό που επετεύχθη στη Μαδρίτη στον τετραμερή διάλογο για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ο δε κύριος Μπρόκ ε, είναι πρόσωπο κλειδί στη διαπραγμάτευση και θα ήθελα να πω πως εκ μέρους της υποεπιτροπής μας είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα και στο επίπεδο των αντιπροσωπιών και στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης. Γνωρίζουμε πως ο συμβασμός περιέχει σαφείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε γενικότερες γραμμές χαιρόμαστε για το ότι το Κοινοβούλιο πέτυχε σημαντικά πράγματα όσον αφορά τη διαφάνεια και την λογοδοσία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το ότι οι προσπάθειες της Επιτροπής μας για πρόσβαση στα έγγραφα αντικατοπτρίζονται στην τελική δήλωση. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριος Μπρόκ να εξηγήσει το συμβιβασμό Να ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μου δίνετε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ε, τα είχαμε συζητήσει ήδη, είναι πράγματι ο συμβασμός αυτός προέκυψε ικανοποιητικό στα βασικά ζητήματα, ίσως η διατύπωση να μην είναι τόσο καλή, αλλά είναι ένα συμβασμό μεταξύ τεσσάρων μερών θεσμικών οργάνων εντό εισαγωγικών και ε, έτσι είναι οι συμβιβασμοί. Αλλά διαπιστώνουμε στα τέσσερα σημεία που σας ενδιαφέρουν και ειδικά στα ανθρώπινα δικαιώματα είχαμε πρόοδο οπότε νομίζω τώρα μπορούμε να ολοκληρώσουμε θα έχουμε μια υπηρεσία η οποία θα ενισχύσει τη δυνατότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν ε, στελεχωθεί σωστά αν έχει τη σωστή ηγεσία και αν αυτά που έχουμε θεωρητικά γίνουν και στην πράξη Δεύτερον, ε, κοινοτική μέθοδος διασφαλίζεται. Λέγεται αυτό παντού πως θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την ΚΕΠΑ και λέγεται πως εκεί που δεν έχει αλλάξει η κοινοτική ε, ευθύνη θα έχει την ευθύνη η Κομισιόν. Δηλαδή όλο αυτό, όλος ο επιχειρησιακός προπολογισμό είναι προπολογισμό Κομισιόν. Οπότε υπάρχει εγγύηση της κοινωτικής μεθόδου. Προγραμματισμός για την πολιτική γειτονία, αναπτυξιακή πολιτική. Μερικά κομμάτια του μέσου σταθερότητα, του μέσου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ευθύνη εκεί είτε αναφέρεται ρητά είτε διαφυλάσσεται. Δηλαδή ότι η ύπατη εκπρόσωπος δρά τότε ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ειδικά αυτό στο τελευταίο κομμάτι της κοινωτικής μεθόδου δεν είναι εύκολο. Και Αυτό το διαπραγματευτήκαμε μέχρι το τελευταίο, το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο μέρος. Δεν είναι δηλαδή, δεν θα υπάρξει μια υφέρπουσα διακυβερνητικοποίηση και βλέπουμε πως θα υπάρξει εδώ πέρα μια κάποια υποχρέωση. Επίσης τα δικαιώματα προϋπολογισμού και απαλλαγής ενισχύονται όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Δεν πρέπει να εγκριθεί δηλαδή μόνο ο προϋπολογισμός, αλλά ό,τι έχει φύγει από το Συμβούλιο και πάει στην υπηρεσία αυτή, μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε μέσω του διοικητικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Όπως κάνουμε με τον προπολογισμό της Κομισιόν. Έτσι ώστε και εδώ υπάρχει έλεγχος ε, κοινοβουλευτικός. Βεβαίως αν πάμε στην ΚΕΠΑ που είναι η υπόθεση του Συμβουλίου έχει γίνει μια συμφωνία κυρίων να έχει περιορισμένα δικαιώματα το Κοινοβούλιο. Για να δούμε τι γίνεται με τις αποστολές ΚΕΠΑ. Πρέπει να είναι διαρθρωμένος ο υπερπολογισμός με λεπτομέρειες, με γραμμές, π.χ. τι γίνεται στο Αφγανιστάν. Ποια είναι η στρατιωτικό κομμάτι, τι είναι το πολιτικό κομμάτι, τι είναι αναπτυξιακή βοήθεια. Και αυτό είναι οπωσδήποτε ενδιαφέρον. και για την πολιτική μας δουλειά και για τη δουλειά του δημοσιονομικού ελέγχου. Επίση, τα ανθρώπινα δικαιώματα καμιά φορά είναι στον τομέα τη ΚΕΠΑ, αλλά υπάρχει εδώ η δήλωση πω η ύπατη εκπρόσωπο υπογράφει πω όχι μόνο σε ζητήματα προπολογισμού, αλλά σε όλα τα ζητήματα η Επιτροπή του Κοινοβουλίου θα έχει δικαιώματα διαβούλευσης πριν ληφθεί η απόφαση στο Συμβούλιο. Δηλαδή, μπορεί εδώ πέρα να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες της για να γίνουν συζητήσεις εκ των προτέρων και να το εξετάσουμε αυτό υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τελευταίο, κυρία Πρόεδρε, γνωρίζετε πως η υπατή εκπρόσωπος λέει πως κάθε πρέσβης είναι και εκπρόσωπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό φαίνεται γιατί υπάρχει κομμάτι ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υπηρεσία αυτή για να μπορεί να έχει και λόγο και αυτό θα γίνει. όχι μόνο σε διορισμούς ε, π.χ. το ότι πρέπει να εμφανίζεται ο νέος πρέσβης ενώπιον της Επιτροπής αλλά στο μέλλον το Κοινοβούλιο θα μπορεί να προσκαλεί αυτούς τους ανθρώπους σε συνεδριάσεις Επιτροπής και θα είμαστε σε δυνατότητα όταν μια χώρα είναι σε, κρίση να καλούμε τον αρμόδιο πρέσβη να μας πει τι τρέχει. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Κατά που είχαμε συζητήσει στην αρχή αυτής της διαδικασίας γιατί πρέπει ως κοινοβούλιο να μην κάνουμε μόνο εκθέσεις και ψηφίσματα να φροντίσουμε οι ρήτρε και οι συνθήκες να ελέγχονται να ελέγχονται από την επιχειρησιακή πλευρά δηλαδή ο έλεγχος για το εάν γίνεται κάτι τέτοιο είναι αποφασιστικός και τα δικαιώματα που αποκτά το κοινοβούλιο, οι δομές αύξησαν τις δυνατότητες να γίνει κάτι τέτοιο πιο ε, φυσιολογικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Η εμείς ευχαριστούμε κύριε Μπλοκ και βεβαίως πρέπει και προσωπικά να σας ε, συγχαρώ για τα όσα πετύχατε σε αυτές τις τόσο δύσκολες διαπραγματεύσεις. Δύο ερωτήσεις έχω. Πότε την επόμενη εβδομάδα θα αποφασίσει από αυτό το κοινοβούλιο και τι θα γίνει όσον αφορά την φάση της παρακολούθησης της εφαρμογή όταν ε, ε, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε το τι θα γίνει, πώς θα έχουμε την πιο δόκιμη συνέχεια. Και επίσης για πέστε μας όσον αφορά την διοργανική συμφωνία και την προσβασιμότητα εκ μέρους ε, του Κοινοβουλίου ή στις πληροφορίες, πώς θα μπορέσετε να λάβετε υπόψη τα όσα πρεσβεύουν οι επιτροπές, οι υποεπιτροπές, κυρίως εμείς, ούτως ώστε να λάβετε υπόψη τι γίνεται όσον αφορά ε, ε, το, το διαμορφούμενο τοπίο. Και να δούμε τι διαστάσεις θα δώσουμε στις προσπαθειές μας. Βέβαια ε, να δούμε και τι θα γίνει με τη Διοργανική Συμφωνία, τι σχετικές διαπραγματεύσει τώρα. Ε, αν θέλετε απαντήστε και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο τους συναδέλφους. Αυτή τη στιγμή το συζητάει η διάσκεψη των Πρόεδρων. Η διαδικασία είναι ως εξής. Μέχρι Δευτέρα το βράδυ θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί η υπηρεσία έτσι ώστε τρίτη πρωί να εγκρίνει την έκθεση η Επιτροπή Εξωτερικών να συζητηθεί την Τετάρτη στις και να ψηφιστεί την Πέμπτη. Το αν θα ψηφίσουμε τώρα την Πέμπτη, ε, δεν ξέρω, οι, οι απόψεις διαφέρουν. Για μένα σημαντικό είναι να έχουμε μια απόφαση και Τετάρτη να γίνει η συζήτηση για να σταθεροποιηθεί και η απάντησή μας στην κυρία Άστον. Τώρα το αν θα προλάβουμε να ψήσουμε ή όχι, εντάξει δεν έχει τραγική σημασία αλλά είναι αρκετά σημαντικό. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε για το τι γίνεται με τον κανονισμό υπηρεσιακής ε, κατάστασης. Θα πρέπει λοιπόν Σεπτέμβρη να δούμε οι αρχές Οκτωβρίου τι γίνεται τι είναι εφικτό. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να γίνει τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης όταν το Συμβούλιο λάβει την απόφαση στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαβούλευσης. Αν δεν τηρήσει τη συμφωνία το Συμβούλιο και φρενάρει ξανά τη διαδικασία, ή φρενάρει τον χρηματοδοτικό κανονισμό ή το ότι θα μπορούν να εξομοιώνουν οι εθνικοί διπλωμάτες με το άλλο προσωπικό εμείς θα έχουμε έτσι την δυνατότητα να μην μας ε, ξεγελάσει θα έλεγα το Συμβούλιο να έχουμε μια διασφάλιση γιατί οπωσδήποτε θα διηγηθούμε σε δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή θα πρέπει να μας απασχολήσει και να το μοιράσουμε. Δηλαδή πρέπει να δούμε την ουσιαστική εφαρμογή που ανήκει στην Επιτροπή, που Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και υπάρχει και ο έλεγχος του προπολογισμού. Και να δούμε πώς θα συνεννοηθούν αυτές οι επιτροπές. Για να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό χαρτί του Κοινοβουλίου για να τηρήσει η Κομισιόν και το Συμβούλιο τα συμφωνημένα. Αλλά νομίζω καλό θα ήταν να πούμε πως αρχή του επομένου έτους να μαζευτούν εδώ πέρα εκπρόσωποι αφού έχει λειτουργήσει μισό χρόνο η υπηρεσία και να δούμε τι έχει γίνει. Και το θέμα της πληροφόρησης μας έχουν υποσχεθεί βεβαίως αυτή την πενταμελή επιτροπή που θα έχει πρόσβαση στα διαβαθμισμένα έγγραφα. Αλλά το πιο ενδιαφέρον για σας. Οι εισηγητές στις επιτροπές αν κάποιος ε, ε, εδώ η Επιτροπή σας βεβαίως πάγεται στην Επιτροπή Εξωτερικών. Οπότε ο πρόεδρος της ΑΦΕΤ μπορεί να απευθύνει επιστολή ή ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στην κυρία Άστον για να δει έγγραφα για να μπορέσει να συντάξει την έκθεσή του ή την έκθεσή του. Π.χ. για τα Αφγανιστάν, ξέρω εγώ. Το άτομο αυτό λοιπόν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δει εμπιστευτικέ πληροφορίε για να γίνει σωστή έκθεση. Και εκεί πέρα είπαμε πως αυτό θα γίνεται είτε με επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών ή του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Äh, να μην ζητάει ο καθένας ε, ό,τι θέλει, γιατί αλλιώς θα μας πούνε ότι δεν λειτουργεί το σύστημα κτλ. Γιατί να υπάρχει, ξέρετε, τα έγγραφα έχουν πάνω και βαθμό ασφαλείας κτλ. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Οπότε θα πρέπει και να συνεργαστεί αυτός ο άνθρωπος με άλλους πέντε μετά στην ε, Επιτροπή. Um, um, Σημειώσαμε τα του νέου μηχανισμού Πράγματι υπάρχει το θέμα των εγγράφων το οποίο περιορίζεται στην ΚΕΠΑ. Ίσως όμως κάποια άλλα έγγραφα απτονται διαφορετικών διαδικασιών και υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες πρόσβασης σε αυτά, ιδιαίτερα για τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε κατά περίπτωση. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες, υπάρχει επίσης και η διοργανική συμφωνία και υπάρχει μια εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου εκεί όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Έχουν γίνει στο παρελθόν κάποιες συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους κανόνες διαφάνειας. Οι συζητήσεις αυτές δεν είχαν καταλήξει κάπου, αλλά υπάρχει επίσης και το θέμα κάποια από τα έγγραφα αυτά για να τα δουν οι βουλευτές να έχουν την δυνατότητα από τη χώρα τους να έχουν αυτή την άδεια αν θέλετε την δυνατότητα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπρόκ, λέει η κυρία Γκόμες, γιατί έχει κάνει πράγματι πάρα πολλή δουλειά. Αυτό το οποίο βλέπω πάντως εγώ εδώ είναι ότι στο έγγραφο δεν δίνεται η δυνατότητα να υπάρξει εποπτεία από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Προηγουμένως συζητούσαμε για το Κονγκό σαν παράδειγμα και η ΜΚΟ διαμαρτυρόντουσαν ότι δεν παίρνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα και εμείς ξοδεύουμε τόσα χρήματα στο Περιφερειακό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή λέει, Επιτροπή λέει ότι χρηματοδοτεί πάρα πολλές οργανώσεις ΜΚΟ κτλ. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το ΦΕΝΤ λοιπόν εδώ και εμείς προσπαθήσαμε να πιέσουμε στην αρχή έτσι ώστε να ενταχθεί στις κανονικές διαδικασίες το ΦΕΝΤ, αλλά αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Πού βρισκόμαστε, δεν ρωτώ με σήμερα. Υπάρχει η δυνατότητα να μη συνεχιστεί η κατάσταση αυτή και να ελέγξει το Κοινοβούλιο. Ναι, αυτό, αυτή η κατάσταση οφείλεται στη συνθήκη της Λισαβόνας, εκεί την πατήσαμε. Αυτό αποκλείεται από την ίδια τη συνθήκη και σχετίζεται με το ότι το μέσο αυτό, το αναπτυξιακό ταμείο, χρηματοδοτείται και διαφορετικά. Εκπροσωπούνται αλλιώς τα κρατημέλη, με άλλη ποσόστοση από την συνήθι ποσόστοση των συνεισφορών γιατί οι πρώην ε, απικιακές δυνάμεις ε, πληρώνουν περισσότερα από ό,τι οι υπόλοιπες και πράγματι αυτό είναι ένα από τα δύσκολα σημεία. Και δεν ε, τα καταφέραμε ε, πράγματι σε αυτόν τον τομέα να έχουμε ε, σαφήνεια στον προϋπολογισμό. Εκεί όμως όπου απαιτείται νομοθεσία, εκεί μπορούμε να εφαρμόσουμε τη συναπόφαση. Αυτό είναι δυνατόν και νομίζω πως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα γενικά μέσα για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και πρέπει να πω πως όταν όλα αυτά τελειώσουν θα πρέπει να πω στην είπατε εκπρόσωπο πως ε, δεν αντιλαμβάνομαι αυτό το διαχωρισμό εγώ δηλαδή πότε δράω ως αντιπρόεδρος και πότε ως είπατε εκπρόσωπος και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην γίνεται διάκριση από πλευράς του ελέγχου δηλαδή και θεωρώ πως με τη μέθοδο αυτή θα βάλουμε έτσι λίγο πόδι στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής Γιατί διαπιστώνουμε βέβαια στο θεσμικό το, το πρόβλημα. Ευχαριστώ τον λόγο έχει κυρία Φάιντερ. Ευχαριστώ πραγματικά για αυτό το οποίο έχει κάνει ο Ολμαρ Μπρόκ. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφορά τις εθνικές ε, ποσοστώσεις στην υπηρεσία γνωρίζω πως κάποιες κυβερνήσεις και οι μικρότερες ε, των νεότερων και μικρότερων κρατών μελών ανησυχούν για το τι γίνεται για την κυριαρχία δηλαδή των μεγάλων και εμπειρών χωρών πως έχει τώρα λοιπόν η κατάσταση των διαπραγματεύσεων και πως θα είναι τα πράγματα και μπορούμε να πιστέψουμε πως οι νέες και μικρές χώρες ε, θα εκπροσωπούνται. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ευχαριστώ. Κύριε Μπρόκ. Δεν, δεν ανέφερε τίποτα στην πρώτη πρόταση άστον. Μετά από πίεση του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών έγινε μια αλλαγή στη θέση του Συμβουλίου όπου μιλάμε για ισορροπία φύλων και γεωγραφική ισορροπία. Επιτύχαμε λοιπόν κάποια πράγματα παραπάνω και άρα περισσότερα από αυτά τα οποία επέτυχαν τα κράτη-μέλη παρά όλο το βέτο που είχαν τα κράτη-μέλη και γνωρίζω τη συζήτηση που λαμβάνει χώρα. Δεν ξέρω τώρα εάν δικό μου καθήκον ήταν να έχω εγώ καλύτερα αποτελέσματα από τους υπουργού εξωτερικών που είχαν και βέτο, υπενθυμίζω. Ε, να είμαστε έτσι και λίγο λογικοί. Τι έχουμε λοιπόν τώρα. Αναφέρεται πως ε, πρέπει να επιτευχθεί η ισορροπία γεωγραφική και των φύλων και αυτό είναι νομικά δεσμευτικό. Αναφέρεται ως στόχος, δηλαδή στα, στο, στο διατακτικό. Είναι δεσμευτικό. Yeah. Πώς να το πω. Και στα εκτιμώντας αναφέρεται πως παραδείγματος χάρη γεωγραφική ισορροπία ισχύει ειδικά για τα κράτη-μέλη τα οποία υποεκπροσωπούνται και πρέπει να ενισχυθεί και επιπλέον λέγεται πως εάν διαπιστωθεί το 2013 πως εξακολουθεί να υπάρχει ανισορροπία τότε θα έχουμε πρόσθετα, πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανισότητα. Ε, νομίζω πως είναι αρκετά. δεν αναφέρει αυτό το οποίο ήθελε ο κύριος Σάρις Βόλσκι περί δικαιώματος συμβουλίου δεν θυμάμαι το νούμερο γιατί ούτως ή άλλως είναι εκτός ισχύως δεν μπορώ εγώ να αναφερθώ γιατί η οδηγία πλέον δεν ισχύει ρωτήστε ένα δικηγόρο Εκείνη η διαφορά. Και δεν είμαι διατεθειμένος να μπω σε εγώ στον ανταγωνισμό αυτό των, και τις διαπραγματεύσεις των, των πρώτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Που ήρθατε εδώ για να μας εξηγήσετε τι ισχύει και ελπίζουμε ότι την επομένη εβδομάδα που θα μπορέσει να έρθει εδώ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και εμείς τι γίνεται με την ε, εφαρμογή όλων αυτών που προβλέπονται και υπό επιτροπή πώς θα μπορέσει να προωθήσει τα τίματά της. Συνάδελφοι, είμαστε τώρα στο 7 στα διάφορα και έχω τον πειρασμό να ζητήσω από τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Μακμίλαν Σκότ, ο οποίος παρίσταται να μας πει για ένα τρίλεπτο τι έγινε ή στην ε, συνάντηση την, ε, των δύο πλευρών του, του, του Ατλαντικού που εκπροσώπη τον πρόεδρο Μπούζε για τη δημοκρατία. Έχουμε, έχουμε λίγα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το είπα πριν στην γραμματεία ότι δεν μπόρεσα να παραστώ σε εκείνη την ε, συνάντηση της Washington. Διότι διότι ε, πέθανε κάποιος συνάδελφος ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν μπόρεσα να πάω. Έγινε σύμφωνα με τα όσο προβλέπει ο οίκος Τσέιθαμ και, και την συνεργασία με τη ΣΥΠΑ όσον αφορά την ε, πρόθεση της δημοκρατίας αυτός ήταν ο σκοπός. Ο κύριος Μπούζεκ πήγε Γιάννα Γκόμες ήθελε να πάρει να πήγε τελικά, αλλά νομίζω ότι θα ενδιέφερε την υποεπιτροπή μας σε μια συνάντηση στο μέλλον να συζητήσουμε για την συνάντηση της Washington. Γιατί και εσείς αποφασίσατε Έχουμε φτάσει στο Ευρύ, επομένω. Τη συνάντηση εκείνη. Στις 13 Σεπτεμβρίου έχουμε την ημέρα ε, της δημοκρατίας. Οπότε θα πρέπει ίσως αυτό να το λάβουμε υπόψη για τις ημερήσεις διατάξεις μας, για τις συνεδριάσεις μας. Γιατί όπως σας είπα δεν μπόρεσα να παραστώ στη συνάντηση. Όμως πήγαν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι και ο πρόεδρός μας. Α, ε, περιεκτική πλήρηση ενημέρωση μας κάνατε, οπότε θα πρέπει όσο γίνεται καλύτερα να, παρακολουθήσουμε το τι θα γίνει για τη δημοκρατία και με μεγάλη μου χαρά α, ε, α, ε, ακούω ότι ο κύριος Μπρόκ ενημερώθηκε γιατί είναι ο πρόεδρος της σχετικής ε, επιτροπής για τον διάλογο με τις ΕΠΑ. Σήμερα το πρωί τα συζητήσαμε κύριε Μπρόκ και ίσως για το διάλογο των νομοθετών θα πρέπει να ληφθεί αυτό μια που έχουμε τέτοια σύγκληση τέτοια ομοφωνία ενότητα μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό να έχουμε αυτό το feedback να έχουμε την αντίδραση, την ανταπόκριση ε, των, των ε, ομολόγων μας της Αλληπλωρός του Ατλαντικού σας ευχαριστώ Κύριε Μπρόκ, ναι. Δεν ξέρω αν θα, θα λάβετε μέρος κι εσείς ε, την ερχόμενη πέμπτη που θέμε να συνεννοηθούμε με τους ε, αντιπροέδρους και την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ για το πώς ε, θα οργανωθούμε. Έχουμε μια σειρά ταξιδιών, δεν είχαμε κάνει συνεννοήσεις και τρελάθηκαν οι Αμερικάνοι γιατί ο καθένας ήθελε να δει τους ίδιους ανθρώπους και υπήρχαν κάποιες δυσκολίες. Άλλη φορά θέμε να συνεννοούμαστε με το γραφείο μας στην Ουάσιγκτον και νομίζω πως αυτό σας ενδιαφέρει και εσάς και τους ε, συναδέλφους και τους συναδέλφους στο Κογκρέσο να έχουμε, ένα, να έχουμε συστηματικές επαφές. Δεν ξέρω. Δηλαδή κάποιοι συγκεκριμένοι να είναι σε επαφή μόνιμη με τους Αμερικάνους. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν θέμε να, να συνεννοηθούμε. Οπότε μπορείτε να έρθετε κι εσείς. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Είναι μια καλή στιγμή αυτή, μια καλή σύμπτωση. Θα πρέπει να τελειώσουμε εδώ. Η επόμενη συνάντηση που είναι η τελευταία πριν από τις διακοπές θα γίνει στις 15 Ιουλίου. Στο επανειδήν.